Ας ξεκινήσουμε. Δευτεριάτικα, ξέρετε, με τις αφήξεις και λοιπά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έχουμε σημαντικά θέματα, φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Δύο αλλαγές έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Μπορείτε να με ακούσετε. Μία είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Αύριο το απόγευμα στις 3, αντί συζήτηση η γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γυναικών της Επιτροπής ΔΕΒ θα γίνεται αλλαγή απόψεων για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Συρία. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Συρία, στο Χαλέπι, βλέπετε σκηνέ και δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατε, εκπρόσωπο κυβερνήσει για να περάσει βοήθεια προ το Συριακό λαό. Και συζητάμε και θα μα πούν τι κάνουν, πόσο επιτυχή υπήρξαμε, ποια είναι τα προβλήματα στο Χαλέπι, η φραγμή. Αύριο το απόγευμα στι μετά από αυτά που συνέβη στην ΑΕΤ το Σαββατοκύριακο, θα αναφερθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια για την ΑΕΤ. Ε, λοιπόν, αν οι βοηθοί μπορούν να ενημερώσουν τα μέλη, να τους πούνε ότι αύριο στις το απόγευμα έχουμε σημαντικό θέμα. Και αν όλοι συμφωνείτε, το προσθέσουμε στην ημερήσια διαταξή. Μείο 10, κάτω από του εισηγητού ΔΕΒ, του Ιγνάθιο Κοράο, εισηγητού γνωμοδότης, να αναβληθεί ψηφοφορία για την πρόσβαση στα φάρμακα, του σημείο 10, να αναβληθεί η ψηφοφορία για να έχουμε περισσότερο χρόνο για σωστή προετοιμασία. Συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω κάποιους Αύριο το πρωί. Να σας υπενθυμίσω. Στις 10. Ψηφοφορία σε 9. Στις 10 μετά. Στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Θα πάμε εκεί Έχουμε δύο κοινά θέματα που συζήτησε με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Το πρώτο, Ευρωπαϊκή εκδήλωση για την Ολέα, να μιλήσουμε στους νέους για τη μεταναστευτική κρίση. Κάθε πολιτική ομάδα έπρεπε να διορίσει ένα μέλος να παρακολουθεί στη διαδικασία. Ελπίζω αυτό να συνέβη. Δεύτερον, κοινή συζήτηση για τις μετακινήσεις ε, των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στις 11.30 ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ. Θα πάμε από εδώ, θα πάμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, στο άλλο κτίριο, στο 2Q2, αύριο το πρωί. Αυτά. Σας υπενθυμίζω τι γίνεται την Τρίτη. Τετάρτη. 9 με 10 και μισή. Κοινή συζήτηση. Με την Επιτροπή δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά στην Αιθιοπία. Είχαμε αναφορές επιθέσεων που συνέβησαν στην Αιθιοπία και θα συζητηθεί από 9 μέχρι μισή Τετάρτη το θέμα αυτό. Και άλλα δύο σημεία, Τετάρτη απόγευμα. Το πρώτο, κοινή συνεδρίαση στις τρεις επιτροπών με την Επιτροπή Περιβάλλον και την Επιτροπή ανάπτυξη. Αλλαγή του κλίματος και αλλαγή καλλιεργιών και τροφίμων είναι για την ημερίδα την Παγκόσμια ημέρα Τροφίμων ε, από τις 3 μέχρι τις 4, την Δετάρτη. 3 με 4 την Δετάρτη. Ταυτόχρονα έχουν προσκληθεί τα μέλη στην Επιτροπή Ίντε, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εκεί υπάρχει ακρόαση 3 με 5 για εμπορική πολιτική και βιωσιμότητα της άγριας πανίδας στην 3G3. Πέμπτη πρωί, περίπου 11.30, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα έχει μια παρουσίαση ειδική εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου. Θέμα ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. διάφορες σημαντικές συζητήσεις επιτροπές. Θα στείλει υπενθύμη στα μέλη γραμματεία με σειρά γιατί δεν έφτασαν και πολλά μέλη, να σα υπενθυμίσει η γραμματεία όλε αυτέ τις εκδηλώσει και τι συζητήσει. Να πω μερικά λόγια για το βραβείο Ζαχάροφ και ψηφοφορία. Λοιπόν, θα, και κλεισμό των θυρών με, στη 2Q2, 11 και 30 γίνει ψηφοφορία και κλεισμό των θυρών και μυστική ψηφοφορία. Κάθε ομάδα μέχρι 6 το απόγευμα σήμερα να μα πει ποιο θα είναι ενδεχομένω αναπληρωτή τη επιτροπή. που θα συμμετάσχει η ψηφοφορία. Πρέπει να συνεργαστείτε και να συντονιστείτε με τα μέλη τη Επιτροπή ΑΦΕΤ. Μόνο οι καταγεγραμμένοι θα μπορούν να λάβουν μέρο στη μυστική ψηφοφορία. Δεν εμφανιστεί κανεί τελευταία στιγμή 11.30 να ψηφίσει. Στείλτε τι πληροφορίε λοιπόν τη κατάλληλη γραμματεία μέχρι τι 6 σήμερα το απόγευμα. Ερωτήσει περί των ανακοινώσεων. Υπήρχαν πολλά που είπα, θα σα στείλουμε μέσω κειμένου. Σημείο 3. Τον Έγκριση πρακτικών. 20 και 21 Ιουνίου. 30 20 Ιουνίου, 11-12 Ιουλίου. Έχετε στο χαρτοφύλακά σας, αν έχετε σχόλια. Κοινοποιήστε τα σχόλια στη γραμματεία πεντός συνεδριάσεως. Άνευ σχολείων θεωρούνται τα πρακτικά ως εγκεκριμένα. Σημείο 4. Και για τη συνεδρίαση των συντονιστών για τα πρακτικά συστάσεις για τις 7 Σεπτεμβρίου, σχόλια στη γραμματεία πριν το τέλος της συνεδριάσεως άνευ σχολείων θεωρούνται και αυτά τα πρακτικά εγκεκριμένα. Σημείο 5. Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε σχόλια? Έχετε κάτι να μας πείτε. Α, α, εκεί είσαστε. Όχι. Τίποτα. Σε αυτό το στάδιο. Ωραία. Ωραία. Κερδίζουμε χρόνο. Σημείο 6 παρακολουθήσει της εφαρμογής των στόχων βιωσίμου αναπτύξεως. Ποιες είναι οι εξελίξεις. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη και δημιουργήθηκε όλη η διαδικασία και ζήτησαν συντονιστές εκπόνηση μελέτης για το πώς εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή για τους στόχους της ε, χιλιετίας. Αρκετοί στόχοι και δείκτες έχουν καθοριστεί. Ζητήθηκε οι κυβερνήσεις να ενημερώσουν και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παραμείνουν νεκρό γράμμα όλα αυτά. Πώς θα τα σχετικά μέτρα. Γι' αυτό ζητήσαμε από, στο, από το τμήμα ερεύνη να ετοιμάσει μια μελέτη. Και αυτή τη μελέτη την έχετε εδώ. Μελέτη που ετοίμασε το Δανέζικο Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών, ανεξάρτητος ερευνητικός φορέας, ο δόκτωρ Νίλ Βέμπστα είναι εδώ που θα παρουσιάσει τη μελέτη. Καθηγητά Webster, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Όπως εξηγήθηκε, το Δανέζικο Ινστιτούτο για Διεθνείς Μελέτες ανέλαβε να αποτιμήσει τα μαθήματα που απορρέουν από την παρακολούθηση υλοποίησεως των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ποια είναι η πρόοδος επιτευχθήσα, ποιες δυνατότητες, ποια τα προβλήματα και να εξετάσουμε και τους στόχους αυτούς καθεαυτούς βιωσίμων αναπτύξεως εν ώψη των, ε, της επαναστάσεως των στοιχείων, όπως αποκαλείται, και να δώσουμε συστάσεις. Πώς να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες αναπτυσσόμενων χωρών να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των στόχων της χιλιετίας. Δύο άτομα εκπονήσαμε την έκθεση, ο υποφαινόμενος και η Έλεν von Η Έλεν Mountwall δεν μπορούσε να παρίσταται εδώ να βοηθήσει στην παρουσίαση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμως να καλύψω και εκείνη. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε το έργο αυτό προσεκτικά. Είναι περιπλοκότατο, πάρα πολύ σύνθετο, λεπτομερέστατο. Τι κάναμε, θέλαμε να δούμε πώς δημιουργείται ευκαιρία μέσω εποπτείας των προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Επιτροπή, να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των στόχων σε όλο τον κόσμο όσον αφορά ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να βασιστούμε σε αποκομιστήσεις εμπειρίες, στα μαθήματα, να δούμε τι στοιχεία έχουμε, ποια είναι τα προβλήματα που μας περιμένουν, τι στοιχεία έχουμε, ποια είναι η μορφή τους και να εντοπίσουμε βασικούς τομείς που θα μπορούσαν να είναι τομείς προτεραιότητας για να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους στόχους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. 10 λεπτά, ένα τέταρτο έχω στη διάθεσή μου. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να δούμε τι γίνεται τη συλλογή στοιχείων στον κόσμο. Εστιαζόμενοι επί των αναπτυσσομένων χωρών. Ήταν και στην εντολή που μα δόθηκε αυτό. Γενικέ προκλήσεις που είναι θεωρητικέ πώ καθορίζεται η φτώχεια, φερρυπίν, το εισόδημα, οι ανισότητες, ε, ανισότητα πλούτου κλπ. Και να, όσον αφορά τα δεδομένα, λείπουν κάποια εκατομμύρια. Έχουμε ακούσει γι' αυτό. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων σε παρόμοιους τομείς να αποκαλυφθεί η ποικιλομορφία και η διαφορά και πώς, ε, σε τι βάθος μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την αποσύνδεση των στοιχείων, από ομαδοποίησή τους. Τέσσερα είδη στοιχείων θα πρέπει να γνωρίζετε αυτά που είναι από τις απογραφές, από τις γενικούς ε, ελέγχους, διοικητικά στοιχεία και ε, διαστημικά χωροταξικά στοιχεία. Τα περισσότερα στοιχεία βασίζονται επί απογραφών και εκθέσεων. Δεν γίνεται συχνά στο Μιανμάρ. Έγινε απογραφή μετά από πολλά χρόνια και αποκάλυψε ότι ο πληθυσμός ήταν 10 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που θεωρούσε η κυβέρνηση και σχεδίαζε βάσει αυτών. Είχαν πέσει έξω 10 εκατομμύρια. Αυτά ήταν από απογραφή, από έρευνε, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Με αυτά τα στοιχεία που ενημερώνουν για τα στοιχεία των απογραφών να μπουν σε μεγαλύτερο βάθο, να καταλάβουμε τι ακριβώ γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο, πέρα από το εθνικό. Διοικητικά στοιχεία. Εγώ είμαι Δεν έχουμε απογραφή. Τα πάντα συλλέγονται μονίμως συνεχώς. Είναι διοικητικά στοιχεία σε ύψιστο επίπεδο, τα οποία παράγουν τα στοιχεία. Είτε μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες, είτε μιλάμε για παραγωγικούς τομείς, γεωργία κλπ. Και γεωδιαστημικά στοιχεία και χωροταξικά στοιχεία. Και εδώ είναι η επανάσταση των στοιχείων. Γίνονται έρευνες και καταχωρούνται όσον αφορά τα στίγματα του GPS συλλέγονται δορυφορικά στοιχεία, συνδυάζονται και με στοιχεία από έρευνε για τη γεωργία Φερρυπίν. Είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία. Διότι ένα από του βασικού τομεί παρεμβάσεω είναι ο εξή. Θε το καλύτερο είδο στοιχείων ή πρόθεσμα βολεύεσαι με αυτό που έχει. Παίρνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προσπαθεί να τα βελτιώσει. Όπω απογραφή και έρευνε. Προσπαθούμε στην έκθεση να τα εξετάσουμε αυτά να δούμε τι μας δίνουν τα στοιχεία, ποια μορφή έχουν, ποιοι είναι οι συνδυασμοί αυτών, όπως ε, γεωχωροταξικά στοιχεία, έρευνες, στοιχεία από έρευνες, πώς συλλέγονται τα στοιχεία. Αν δείτε λοιπόν, εδώ έχουμε ένα χάρτη. Μάλλον πρωτόγονος, αλλά χάρτης είναι. Στη σελίδα, σελίδα 11. Μας δείχνει ο χάρτης, είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και δείχνει τη δυνατότητα συλλογή στοιχείων για την ώρα. όπω βλέπετε, για μεγάλο κομμάτι τη Αφρική αυτή η δυνατότητα είναι πολύ μικρή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αναφέρουμε και στις συστάσεις μας. Επίσης βλέπουμε και την αλλαγή από τους στόχους ηλιετίας προς τους, βιώσιμους, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και αναφέρουμε διάφορα συγκεκριμένα σημαντικά στοιχεία από αυτού. Πάμε από 8 σε 17 στόχους και από 60 σε 130 δείκτες. Αρκετά δραματική η αύξηση. Πολλά καλά μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για τη χιλιετία και έχουμε συλλέξει πολλά καλά στοιχεία λόγω των λογοστόχων. Αλλά τι λέμε, ότι τα περισσότερα στοιχεία αφορούν τους τομείς των στόχων της χιλιετίας, κυρίως κοινωνικό τομέα, παιδεία και υγεία, φτώχεια. Υπάρχουν και άλλοι τομείς όσον αφορά τους στόχους της χιλιετίας. Παραγωγή, φυσικούς πόρους, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά κενά όσον αφορά τα στοιχεία, σημαντικά κενά. Όχι μόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και σε χώρες μεσαίου εισοδήματος και καμιά φορά και σε χώρες που είναι πλούσιες. Έχουμε πολλά κενά στα στοιχεία διότι οι στόχοι της χιλιετίας καλύπτουν πολύ ευρύτερο φάσμα στόχων και ευρύτερο φάσμα δικτών. Δεν είναι μόνο το εύρος των δικτών που είναι το πρόβλημα για στόχους χιλιετίας, αλλά και το βάθος αυτών. Διότι οι στόχοι της χιλιετίας εργάζονται με μέσους όρους. Εδράζονται επί μέσων όρων, μέση, μέσος όρος υγείας, μέσους όρος παιδείας κλπ. Οι στόχοι της χιλιετίας αυτή καθεαυτή απαιτούν να μπει κάποιος σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Ταυτότητα, τόπος, ηλικία, εθνότητα. Εσωτερική αξιολόγηση πρόοδου δηλαδή, που είναι κάτι καινοφανές όσον αφορά τους στόχους της χιλιετίας. Τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τους στόχους χιλιετίας και δεν έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες για τη συλλογή αυτού του είδους των στοιχεία. Να δούμε κατά πόσο σε ένα συγκεκριμένο τόπο ορεινό στο Νεπάλ, ε, πετυχάνουν την ίδια πρόοδο όπως στην κοιλάδα του Κατμαντού. Ένα παράδειγμα. Και άλλη σημαντικότατη διαφορά. Αυτή η στόχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι παγκοσμίω εμβολία, συγγνώμη. Δεν αφορά μόνο τις όμνες χώρες. Αυτοί οι στόχοι θεωρούνται Θεωρείται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζονται από τι ανεπτυγμένες χώρες μέσω διεθνών συστημάτων ε, ενίσχυσης για να παρακολουθείτε και η πρόοδο προ την επιτυχία των στόχων. Ισχύουν οι στόχοι για όλες τις ε, χώρες που έχουν υπογράψει. Αυτό αναφέρθηκε, που έχουν υπογράψει στη Νέα Υόρκη. Έχουμε ένα στοιχείο αριθμητικό στη σελίδα 19. πίνακα 4, ω στοιχείο 4. Είναι λίγο περίπλοκο. Δείχνει σαφώ όμω εκεί, ανάλογα με κάθε στόχο, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για δείκτες. Τι δείχνει εδώ. Σε ιδεώδη κατάσταση, όλες αυτές οι γραμμές θα ήταν πράσινες. Θα υπήρχαν επαρκή στοιχεία για κάθε δείκτη για συγκεκριμένο στόχο, για να γίνει σωστή αποτίμηση της επίτευξης του στόχου. Όπως βλέπετε, για τους περισσότερους δείκτες δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέγαμε. Τα τρία επίπεδα. Κατά πόσο είναι ισχυρά τα στοιχεία, λιγότερο ισχυρά ή αδύναμα. Τρία επίπεδα. Τι βλέπουμε εδώ, ότι έχουν πολύ δρόμο μπροστά μας. Όχι μόνο στις χώρες χαμηλών εισοδημάτων, αλλά μεσαίου εισοδήματο και σε κάποιες ανεπτυγμένες χώρες. Έχουμε δρόμο να κάνουμε πριν έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορέσουμε να εξεργαστούμε τους συμπεφωνηθέντες δείκτες. Αναφερόμαστε στην επανάσταση των στοιχείων, των δεδομένων και τι δυνατότητε δημιουργούνται από αυτή. Και κυρίως με τα μεγάλα στοιχεία, big data όπω αποκαλούνται. Τεράστιες δυνατότητε έχουμε. Μα αν βελτιώσουμε την υπάρχουσα μορφή στοιχείων μέσω απογραφών, τακτική συλλογή, ταχεία συλλογή αυτών, γίνεται ταχύτερη ανάλυση των στοιχείων, εκθέσει που συλλέγονται όχι επί χάρτου αλλά σε ηλεκτρονικές συσκευές και και που διαβάζονται άμεσα και γίνεται ομαδοποίηση των στοιχείων. Άρα υπάρχουν μεγάλα ωφέλη και μπορούμε να προχωρήσουμε, τα αναφέρουμε στο έγγραφο. Καλύτερα στοιχεία, αυξημένη συλλογή στοιχείων, βελτιωμένη ανάλυση καλύτερη βάση για διαμόρφωση πολιτικής και παρακολούθηση υλοποίηση πολιτικών, καλύτερε δυνατότητες για συνδυασμό διαφόρων ειδών στοιχείων. Αλλά όπως αναφέρουμε, αυτό είναι κάτι που απαιτεί νέα πλαίσια για τυποποίηση και έτσι να γίνεται σωστή διαχείριση των στοιχείων και ανάλυση αυτών. Και τα πλαίσια αυτά δεν υπάρχουν ακόμα. Πλαίσια για την προστασία των ατόμων από κατάχρηση στοιχείων πλαίσια για την ενίσχυση της αναλύσεως στοιχείων και την αποφυγή στρεβλώσεως στοιχείων και πολλά περισσότερα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα προς αντιμετώπιση. Απαιτείται επίσης, φέρνοντας τα big data μέσα, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ προχωρημένος για τη συλλογή των σημαντικών στοιχείων big data, αλλά οι συμπράξεις με κυβερνήσεις, με εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όσον αφορά την χρήση των στοιχείων με αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, αυτό χρειάζεται επεξεργασία. Το έγγραφο εξετάζει και τα προβλήματα του αόρατου χαρακτήρα, δηλαδή τα, τα εκατομμύρια που λείπουν Φερρυπίνη. Ανέφερα το Νεπάλ. Είχε, έχει σύστημα με κάστες στο Νεπάλ. Τα πρώτα στοιχεία συνελέγησαν το 90. Πριν από αυτό η κάστα ε, είναι ένα θέμα δηλαδή για να δεις πώς αναπτύσσονται διάφορες κοινωνικές ομάδες και αυτό δεν είχε ληφθεί υπόψη η κάστα. Ε, το ίδιο επίσης στην Ανατολική Αφρική, οι ομάδες Βοσκή και στο Μιανμάρ, στην Αιθιοπία, στην κοιλάδα του Όμο, όπου ε, δεν υπάρχει σωστή καταγραφή των πληθυσμών ανάλογα με εθνικότητα κλπ. Υπάρχει έλλειψη εκατομμυρίων και να όπως σας είπα και τελικά το έγγραφο αναφέρεται στον έλεγχο παρακολούθηση, εποπτεία ε, είναι πολύ σημαντικό για τη λογοδοσία. Και βλέπουμε και την πολιτική βούληση. Συνειδητά και ασυνείδητα υπάρχουν πολιτισμοί και νοοτροπίες που, πώς να το πω, διοικητικές νοοτροπίες που δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία διότι δημιουργούνται νέε μορφέ λογοδοσία. Αυτό χρησιμοποιείται πιο πολύ αποτελεσματικά στη διαχείριση τη τοπική αυτοδιοίκηση μέσω συστημάτων αποτιμήσεω αποδόσεω. Αυτή η λογοδοσία και ο έλεγχο, πώ να το πω, είναι αμφίσιμο τομέα, ε, επίμαχο. Και ίσω εκεί καθυστερήσαμε ε, όσον αφορά τη δημιουργία του κατάλληλου υποπτικού πλαισίου. Κλείνοντα, ε, τι αναφέρουμε. Φύγουμε έξι τομεί, όπου εκεί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκριτικό όφελο. Άρα μπορεί να θέσει προτεραιότητε και να προωθήσει τον έλεγχο τη επιτεύξεω των στόχων μέσω σε συνεργασία με τι αναπτυσσόμενε χώρε, με του εταίρου τι αναπτυσσόμενες χώρε και ευρύτερα, διότι είναι παγκόσμια η φύση των στόχων. Πρώτα απ' όλα, η απομαδοποίηση, ο διαχωρισμό των στοιχείων αύξηση της δυνατότητας εντός χωρών να γίνεται σωστός έλεγχος και όχι μεταξύ χωρών. Να απομακρυστούμε από επιδόσεις μέσω όρου σε μια χώρα και να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό για διάφορες εθνοτικές ομάδες, πολιτισμικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, ομάδες βάσει οικονομικών συνθήκων. Έτσι μπορεί κανείς να έχει περισσότερες αποχρώσεις στην εικόνα σχετικά με το πώς προχωρούμε προ την επίτευξη των στόχων. Δεύτερον, όσον αφορά την αλληλουχία εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ε, έχουν μεγάλη ε, έχουν πλονεκτική θέση. Πρώτα απ' όλα αλληλουχία από έλεγχο και απογραφή και στοιχεία σχετικά να πάμε προς τα διοικητικά στοιχεία. Δηλαδή να παράγονται ε, συνεχώς ροές στοιχείων, σταθερές ροές στοιχείων. Να δούμε βραχυπρόθεσμα τι μπορούμε να πετύχουμε και μακροπρόθεσμα τι μπορούμε να πετύχουμε χρειάζεται να εντοπίσουμε την αλληλουχία για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να μετακινηθούμε και να αλλάξουν τα πράγματα. Μετά υπάρχει και άλλη μια δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την αλληλουχία της επένδυσης. Δεν επιτυγχάνονται στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο ρυθμό όλες, όλοι οι στόχοι. Άρα πρέπει να δίδεται η ενίσχυση και η προώθηση με κατάλληλη αλληλουχία Α πούμε εθνικά στατιστικά στοιχεία, πώ μπορούν να παράγονται και να ανλύονται σε βασικού τομεί, εκεί που μπορούμε να πετύχουμε τα περισσότερα κέρδη. Το συζητούμε και αυτό σαν μία από τι προτεραιότητες. Επίσης, αναφέρουμε τη δυνατότητα να συμβάλλεται στην παρακολούθηση των παγκοσμίων οικονομικών χρηματοστοτικών ροών. Η διεθνής οικονομική βοήθεια δεν θα είναι ο πρωταρχικός στόχος στήριξης για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να παρακολουθεί κανείς συνοτοπιστατικές ροές, ιδιωτικές και άλλες ε, και αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Θα αυξανόταν η ροή των πληροφοριών. Οι διάφορες αρχές φορολόγησης ε, θα μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα το τι γίνεται στις χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα. Και το ψηφιακό χάσμα, άλλος κινδύνος. Όχι μόνο σοφά πληροφορίες αλλά και πρόσβαση πληροφορίες και αυτό είναι σημαντικότατο τομέα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ψυχιακές πληροφορίες επεκτείνεται τάχιστα, αλλά επεκτείνεται ταχύτερα για κάποιους από ότι για άλλους. Και υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος κάποιοι να μείνουν πίσω. Και πιο συγκεκριμένα, τομέας του ελέγχου του τι ακριβώς συμβαίνει, πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι, Πώ ετοιμάζονται τα κριτήρια για την παιδεία, πώς επηρεάζονται τα κριτήρια για την παιδεία, τι επενδύσεις κ.ο.κ. Αναφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να είμαστε στην πρώτη γραμμή για τους μηχανισμούς περιφερειακής ε, αναθεώρησης για το πρόγραμμα, το θεματολόγιο του 2020, θεσπίζοντας μηχανισμό περιφερειακού ελέγχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. μπορούμε να ηγηθούμε σε αυτό το τομέα. Τέλος, αναφερόμαστε στη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διαχείριση των στοιχείων, ιδιωτικότητα, δηλαδή όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν στην παρακολούθηση της προόδου και τον έλεγχο και την κατεργασία των στοιχείων. Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, συγκεκριμένες συστάσεις. Σκιαγραφώ τώρα το γενικό πλαίσιο των βασικών θεμάτων που προσπαθήσαμε να καλύψουμε προετοιμάζοντας την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε πολλή συζήτηση στην Επιτροπή εν σχέση με τη σημασία αυτή τη αποσένδεση των στοιχείων και χαιρόμαστε που αναφερθήκατε σε αυτό και ότι ένα από τα προγράμματά μα ε, ε, σχετίζεται με το θέμα τη ισότητα των φύλων. Και αν δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω, θα πρέπει να υπάρξει ένα τρόπο να καταμετρηθεί αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και μας δώσετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες εδώ. Η Heidi Hautala έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε και εσάς για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία ελπίζουμε θα συμβάλλει στη βελτίωση της εφαρμογής των ε, αναπτυξιακών στόχων σε εθνικό επίπεδο. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε να διδαχθούμε κάτι με όρους χρήσης των στοιχείων στην περίοδο εφαρμογής από την εποχή ε, που είχε γίνει η διαπραγμάτευση εν σχέση με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς ε, στόχους. Γιατί ε, πιστεύω ότι αυτό ενδεχομένω έχει κάποιες ε, επιπτώσεις εν σχέση με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των ε, στόχων ε, και κατά πόσο η χρήση αυτών των στοιχείων με έναν διαφορετικό τρόπο θα το αλλάξει αυτό. Δεύτερον, επειδή το θέμα της εφαρμογής δεν αφορά μόνο αυτούς τους εν λόγω στόχους και δείκτες, αλλά αφορά επίσης τον τρόπο με τον οποίο θεσμικά όργανα εργάζονται προς την κατεύθυνση της εφαρμογής. Και γι' αυτό θα ήθελα να σχίσω κάποια πίεση, να μας πείτε το πώς θα μπορούσατε να συμβουλέψετε τα θεσμικά όργανα, ούτω ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με ένα πιο περιεκτικό τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και στο πλαίσιο αυτό να χρησιμοποιηθούν και τα νέα στοιχεία με τον καινούριο τρόπο Άρα λοιπόν ο όρος εφαρμογή ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κλειδί όσον αφορά την χρήση αυτή των δεδομένων. Κύριε Βέψε, θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, δυσκολεύτηκα κάπως να σας ακούσω, αλλά νομίζω ότι ε, κατάλαβα τις δύο ερωτήσεις που υποβάλατε. Η πρώτη αφορούσε το γεγονός ότι έγινε μια πολύ μακρά ε, περίοδος διαπραγμάτευσης ε, και το ερώτημα ήταν πώς θα περάσουμε από την εποχή της διαπραγμάτευσης στην φάση της εφαρμογής. Και πράγματι αυτό, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, σημαντικό ερώτημα. Και κάναμε αρκετές υποδείξεις, κάναμε αρκετές υποδείξεις στο ίδιο το κείμενο της μελέτης. Αλλά μιλώντας και πέρα από αυτό, ε, θα έλεγα ότι πιστεύω ότι το ζητούμενο είναι να γνωριστούν οι ρεαλιστικοί στόχοι βράχει πρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, σε πολλές χώρες. Και ε, πραγματικά θα ήταν ευκταίο και ίσως αυτό από τη δεύτερη ερώτησή σας θα ήταν πολύ καλό εάν θα μπορούσαν τα διάφορα υπουργεία να μπορούν να συνεργαστούν με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες ή τα αντίστοιχά τους σε διάφορες χώρες ε, μαζί με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, με ένα πιο ολιστικό, περιεκτικό τρόπο όσον αφορά την συλλογή των δεδομένων και την συμπλήρωση διαφόρων τύπων δεδομένων και όπως είπα συμπεριλαμβάνοντας και τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βραχυπρόθεσμα εγώ θα έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό δεν είναι πολύ ρεαλιστικό όσον αφορά την άμεση επίτευξή του. Και πιστεύω ότι ίσως βραχυπρόθεσμα το ζητούμενο θα ήταν να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των δεδομένων τα οποία ήδη έχουν συλλεγεί για παράδειγμα όσον αφορά τι κοινωνικέ υπηρεσίε, την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. τέτοιου είδου τομεί. Και κατά δεύτερον, να επικεντρωθούμε σε ορισμένου από του τομεί κλειδιά όπου υπάρχουν ισχνά δεδομένα, ενώντας με αυτό το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη, τη χρήση της γης, τους φυσικούς πόρους κλπ. Ε, παρά να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους δείκτες ε, και όλους τους 17 ε, εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους. Και εδώ σκέφτομαι βεβαίως και τις αναπτυξιακές ξόμενες χώρες και ίσως βραχυπρόθεσμα θα έπρεπε να επικεντρώσουμε στην ενίσχυση των όσων έχουν ήδη γίνει πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο επικεντρώνοντας σε ορισμένους βασικούς τομείς όπου τα δεδομένα είναι πενιχρά. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να ε, πυροδοτήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της ικανότητας αυτής και ενδεχομένως θα ενίσχυε την αναπτυξιακή συνδρομή η οποία παρέχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μέσω της Επιτροπής και ίσως με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε το μία αλλαγή την οποία έχουμε εμείς κατά νου για το έτος 2019 και έτσι αναφέρουμε στον έγγρα, στο έγγραφο ως βραχυπρόθεσμη προοπτική. Δεν ξέρω αν ε, σας κάλυψα, ίσως είμαι πιο πίσω από τη δική σας ερώτηση, δεν ξέρω. Ωραία λοιπόν. Ξέρω ότι παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας δώσουμε σε λίγο το λόγο. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Δεν ξέρω την Επιτροπή τι προτίθεται να κάνω σαν αφορά το συντονισμό. Δεν ξέρω ε, αν έχουμε και κάποιον από τη Eurostat. Πώς λοιπόν γίνεται ο συντονισμός ε, και κατά πόσο υπάρχουν σχέδια υποστήριξη τη ε, αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, γιατί εκεί υπάρχουν ελλείμματα. Κατά πόσο λοιπόν η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες. Ο Νόρμπερτ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Βέπστερ. Η ομιλία σας ε, κατέστησε σαφές ότι η συγκέντρωση των στοιχείων, η συλλογή στοιχείων είναι αρκετά περιορισμένη. Και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Και είπατε ότι υπάρχουν σε ορισμένου τομεί, ε, υπάρχουν στοιχεία και σε άλλου όχι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι επαρκή, ούτω ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στην ενέργεια, στο καθαρό νερό κλπ γιατί νομίζω ότι στην πράξη το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο είναι απολύτως ακριβή τα στοιχεία, αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι να δούμε τις γενικότερες τάσεις και να καταστήσουμε σαφές ότι μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και ως Επιτροπή, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να σκεφτούμε το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα οποία γίνονται κάθε χρόνο ή δεν γίνονται. Και νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης ε, πραγματικά θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, αλλά και άλλες επιτροπές. Ε, όταν το διακύβευμα είναι η ανισότητα, για παράδειγμα, στην οταν το διακυβευμα ειναι η ισότητα των φύλων, για παράδειγμα εδώ καλείται η Επιτροπή των γυναικών να συμπράξει ή όταν πρόκειται για θέματα του περιβάλλοντος η αντίστοιχη επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό δεν, το μήνυμα δεν έχει φτάσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί συνεχίζουμε να έχουμε την παλαιά αντίληψη ότι θα, για παράδειγμα, η στόχη της είναι αποστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αλλά τώρα υπάρχει ένας νέος προσανατολισμός γιατί η βιώσιμη αναπτυξιακή στόχη είναι πολύ ευρύτερη. Ίσως θα έπρεπε εδώ και η Επιτροπή να μας ε, πει τη δική της θέση. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπάρχουν κενά στα δεδομένα και μας δείξατε και εκεί το γράφημα που έχουμε δεδομένα και που δεν έχουμε. Πόσο καιρό νομίζετε μας χρειαστεί για να βρούμε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθήσουμε να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία και να περιμένουμε μάλλον τη συλλογή των δεδομένων αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο αν θέλουμε να ελοποιήσουμε και τους ε, στόχους βιώσιμης ε, ανάπτυξης, γιατί όπως και να έχει πρέπει να συλλεγούν αυτά τα δεδομένα πριν ολοκληρωθεί η εφαρμογή των στόχων της χιλιατηρίδα. Επομένω, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό και πόσο χρόνο έχουμε, ιδίω ό,τι αφορά τις βιώσιμες ε, χώρε. Θα σα δώσω το λόγο και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Πρώτον, νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά την τυποποίηση. Ενώ αφενός έχουμε καταφέρει πολλά ε, σε συγκεκριμένους τομείς της συλλογής δεδομένων, υπάρχει μία συμφωνία σε ό,τι αφορά την ολογική ε, διάσταση, αλλά και τη μεθοδολογία ως προς τη μέτρηση. Αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχουν αναλάβει αυτή τη στιγμή ε, στην ε, ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα. Στο Μάρτιο, όπως αναφέρουμε, το Μάρτιο, όπως αναφέρουμε και στην έκθεσή μας, βλέπετε ότι αρκετοί από τους δείκτες ε, ήταν της τρίτης κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε συμφωνία επί της μεθοδολογικής προσέγγισης, υπήρχαν πολύ λίγα δεδομένα. Το Σεπτέμβριο η ίδια ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα ως προς ε, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ επανεξέτασε τους ε, δείκτες και είδαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση ε, ως προς τους δείκτες και τα δεδομένα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αυτούς τους δείκτες. Έτσι βλέπουμε ότι κάποια δεδομένα πήγαν από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 1. Για παράδειγμα, τα δεδομένα για τη φτώχεια. Υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικοί τρόποι επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα και έτσι εντελώ διαφορετικέ ε, συστάσει πολιτική. Αυτό δεν επιτυχάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια χρονιά στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει για καιρό και με έντονο τρόπο για να καταφέρουμε να τα λύσουμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί από τα έξω. Είναι προαιρετική η προσέγγιση. Νομίζω αυτή η ορολογία ε, χρησιμοποιείται. Θέλουμε λοιπόν ε, ε, να παροτρύνουμε και τις κυβερνήσεις της χώρες να στηρίξουν την ανάπτυξη μιας πιο τυποποιημένης προσέγγισης αξιοποιώντα και τι εθνικέ του στρατηγικέ για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και ούτω καθεξής. Αυτό συνδέεται και με το δικό σα ερώτημα, γιατί είναι όντω ένα ένα στόχο που θα μας πάρει καιρό. Δεν ξέρω αν θα το έχουμε πετύχει μέχρι το 2030, αλλά σίγουρα θα ε, έχουμε διανύσει μεγάλο τμήμα της απόσταση προ μια συστηματική συλλογή δεδομένων. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο. Ένα θέμα είναι πώς θα φύγουμε από αυτή την κατακαιρματισμένη, ε, αποσπασματική ε, προσέγγιση προς τα δεδομένα. Και συμφωνώ με αυτό που υπονοείται, ότι ενδεχομένω οι προκλήσει τη παρακολούθηση τη συλλογή δεδομένων ε, ω προ του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη ενδέχεται να υπερβαίνει απλώ ε, το θέμα της, ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρέπει πούμε, να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη εμπορική πολιτική ή τη περιβαλλοντική πολιτική της διαχείρισης ε, φυσικών πόρων, τη διακυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αποσπασματική προσέγγιση. Να μην δουλεύουμε δηλαδή πλέον με στεγανά. Ε, μπορεί έτσι να είναι πιο πολύπλοκο το εγχείρημα, όμως μετά η ποιότητα του αποτελέσματος και οι δυνατότητες που μας ε, δίνει για τη συνέχεια είναι πολύ μεγαλύτερες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Νταρότα απάντησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Eurostat δεν ξέρω αν ε, θέλει να πάρει το λόγο. Εντάξει, μόνο εσεί. Δεν το έχω πει εκ των προτέρων, οπότε δεν θέλω να σας θέσω υποπίεση. Όμως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε κατά πόσο θα επαρευρεθείτε τον ή μάλλον αν παρακολουθήσατε την ετήσια έκθεση ε, τον Ιούλιο και τη σχετική συνάντηση ψηλού επίπεδου, αν έχετε πληροφορίες, ε, θα θέλαμε να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει θέμα με, τους, ε, με τα μικρόφωνα αν γίνεται ο τεχνικός ε, να διορθώσει τα μικρόφωνα. Προς το παρόν ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας ε, στο κανάλι 0, γιατί όντως δεν είναι καλός ο ήχος. Εντάξει, προσθέσω να μιλάω πιο δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Εργάζομαι στην μονάδα DEFCO, μια μονάδα πολιτικής. Ασχολούμαι με ζητήματα δεδομένων και δικτών σε ό,τι αφορά την ψηφιακή επανάσταση, μπορώ, ε, μάλλον την ε, επανάσταση προ τα δεδομένα, μπορώ να σα παρουσιάσω αυτά που κάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΤΕΦΚΟ. Ε, βρισκόμαστε συνεχώ σε επαφή με του συναδέλφου από την Eurostat, δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, αλλά συνεχώ συνεργαζόμαστε για ζητήματα τέτοια. Εάν χρειάζεται και άλλε πληροφορίε, για συγκεκριμένα θέματα, μπορώ να σα τα βρω και να σα τα στείλω γραπτό μετά τη συνάντηση. Ω προ τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την ΤΕΦΚΟ και έχουμε συμμετάσχει ε, και στις διαπραγματεύσεις για το θεματολόγιο για το 2030 πρόπερση σε διάφορες θεματικές ενότητες, ιδίως ό,τι αφορά την μέτρηση, την παρακολούθηση και τα δεδομένα. Πάντα εμείς βέβαια θέλουμε και επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σημασία ε, των ε, ανοιχτών προσβάσιμων ποιοτικών και αναλυτικών στοιχείων και χαιρόμαστε που όλα αυτά πολύ έντονα αντικατοπτρίζονται και στην, ε, στο θεματολόγιο της Αντισαβέμπα, αλλά και τώρα στις συνεχιζόμενες εργασίες μας για την ε, αναθεώρηση της ε, συνενετικής πρότασης. Επομένως είναι πολύ σημαντικό. Μαζί με την κύριο θα παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν για την παρακολούθηση και τις μετρήσεις. Ξεκίνησε ως μια ανοιχτή ομάδα εργασία το 2013 και μετά μέσω ε, της διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας και εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε πέρσι. Και τώρα σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση μεταξύ θεσμικών οργάνων και πώ μπορεί να γίνει ο συντονισμό, Υπάρχει συντονισμό και με τη Eurostat αλλά και με τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά γίνονται μέσω του συντονισμού. Σίγουρα προσπαθούμε να μην δουλεύουμε στεγανά, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και προσπαθούμε να τα στείλουμε ε, σε όλες αυτές τις δομές που σας προανέφερα. Βεβαίως γνωρίζουμε αυτό που ανέφερε ο καθηγητής για τις κατηγορίες, ε, αλλά και ε, τις ενημερώσεις που λάβαμε το Σεπτέμβριο. Σίγουρα θα υπάρξουν και νέα στοιχεία με νέες μεθοδολογίες και θα δούμε και πώς θα κλείσουν ορισμένα ε, κενά στα δεδομένα. Όμως το πιο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Μία από τις ε, βασικές προκλήσεις και δυναμίες ε, της μέτρησης ε, στους στόχους της ήταν πώς θα παρακάμψουμε, αν θέλετε, τις εθνικές αρχές. Γιατί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία βρισκόταν στο προσκήνιο και είχε αναλάβει τα ενία, όμως πολλές φορές δεν υπήρχε συντονισμό με την Εθνική Υπηρεσία και έτσι καταλήγαμε σε διαφορετικά δεδομένα. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά διδάγματα που αντλήσαμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των δικτών, την παρακολούθηση των δεδομένων και την παρακολούθηση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα πολιτικής που αναφέρατε στην έκθεσή σας, συμφωνούμε τα διοικητικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά. Ιδίω σε εμά, σε ό,τι αφορά τι βιώσιμε, ε, συγγνώμη, αναπτυσσόμενε χώρε, θέλουμε βιώσιμα στοιχεία, γιατί κάθε χρόνο έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, 15 εκατομμύρια παιδιά που γεννιούνται και δεν καταγράφονται. Αυτό αφορά τα πιστοποιητικά γέννηση, είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι ένα από του τομεί όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί τεράστια ε, πρόοδο πολύ γρήγορα και συνδέεται με τα διοικητικά δεδομένα. Με τα πηγές καλύπτονται πάνω κάτω οι στόχοι όχι τη κριτηρίδα. Εντάξει, ακόμα κάποια πράγματα μένουν να γίνουν, αλλά μετά οικονομική διαδικασία περιβάλλουν και αυτά είναι σημαντικά. Θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν του κλάδου ε, στου οποίου παράγονται αυτά τα δεδομένα. Συμφωνούμε ε, σε ό,τι αφορά την επανάσταση για τα δεδομένα στα ευρωπαϊκά ζητήματα η σα μπορεί να βοηθήσει, αλλά υπάρχει πίεση χρήση των big data σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω και εμεί ενθαρρύνουμε του εταίρου μα να αξιοποιήσουν και να δαμάσουν, αν θέλετε, αυτόν τον νέο τεχνολογικό κλάδο, αλλά ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο το θέμα, υπάρχουν και ζητήματα ε, ιδιωτική σφαίρα ζωή. Ε, υπάρχουν πολλέ προκλήσει και εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και εθνικέ στατιστικέ υπηρεσίε είναι αυτέ που ηγούνται τη διαδικασία. Τους παροτρύνουμε λοιπόν και εμείς είμαστε σε επαφή με τον ιδιωτικό κλάδο. Πρέπει να υπάρχει ε, αμοιβαιότητα και να μην παρακάμπτονται οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. για τη μεθοδολογία. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση ε, και συντονισμό αυτών των μεθοδολογιών για πολλέ χώρε και αυτό μάθαμε και από του τόπου τη Ότι τα κράτη-μέλη κάποιε φορέ ε, χρησιμοποιούσαν διαφορετικέ μεθόδου σε σχέση με του ε, οργανισμού του ΟΗΕ και έτσι είχαμε πολλαπλά σύνολα δεδομένων για τα ίδια ζητήματα κάποιε φορέ. Έχουμε στηρίξει την ε, στατιστική ικανότητα στι αναπτυσσόμενες χώρες εδώ και καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κάποιες φορές αυτό εντάσσεται σε άλλα προγράμματα στήριξης του προπολογισμού, άλλες φορές είναι ξεχωριστά προγράμματα. Ας πούμε τώρα έχουμε ένα παναφρικανικό πρόγραμμα 7 εκατομμύριων ευρώ για τα αφρικανικά στατιστικά συστήματα. Θέλουμε να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Αφρικανικών Στατιστικών Στοιχείων. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σε συνδυασμό με την Eurostat. Έχετε λοιπόν και πάλι αυτή τη συνεκτική προσέγγιση. Και για την αποσύνδεση των στοιχείων, η απομοτοποίηση και εμεί ε, συνεργαζόμαστε με την Διπηρεσιακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και χαιρόμαστε πολύ που συστάθηκε μια ξεχωριστή ομάδα εργασία το Μάρτιο ακριβώ για την αποσύνδεση των δεδομένων. Συμμετέχουμε λοιπόν στις εργασίες, γιατί θεωρούμε ότι αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό τον, την επικεφαλίδα του θεματολογίου, ε, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, τότε χρειαζόμαστε για τέτοια αναλυτικά στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Mm. Θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, να πω μόνο ότι ε, με τα χαράς άκουσα όλα αυτά τα βήματα. Να προσθέσω μία ακόμα διάσταση μόνο Συμφωνούμε απολύτω ότι αφορά την ενίσχυση τη ικανότητα των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και να δούμε πώ αυτό μπορεί να ενισχυθεί και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι πώ αυτό θα ε, μεταφερθεί και στο ε, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Μιλήσατε και για τη διοικητική ικανότητα που είναι ε, μια δυνατότητα που υπάρχει στι περισσότερε χώρε. Όμω, ε, λειτουργεί μάλλον σποραδικά, δεν αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ε, στη συλλογή δεδομένων και δεν χρηματοδοτείται παρκώς. Και μετά η σύνδεση ε, της τοπικής ε, διακυβέρνησης και της εθνικής διακυβέρνησης, η διασύνδεσή τους λοιπόν είναι ε, πολύ χαμηλή στις περισσότερες χώρες χαμηλού εισοδήματος. Όμως όλα αυτά που, που αναφέρατε εσείς ε, εντάσσονται και στην έκθεσή μας. Επομένως, ε, συμφωνούμε απολύτως. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ε, φαίνεται ένα ξερό ζήτημα το θέμα των στατιστικών, όμως... Είναι πιο σημαντικό από αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Επομένως, χαιρόμαστε πολύ για αυτό που είπατε για την Αφρικανική Ένωση και θέλετε να στηρίξετε τη στατιστική υπηρεσία εκεί. Αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλουμε να τα ξανασυζητήσουμε τον Νοέμβριο, μάλλον τον Νοέμβριο, και με τον εισηγητή μας για την υλοποίηση των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Το συναντήσαμε και ε, προηγουμένως και μας μίλησε για τη σημασία αυτού του έργου που συνεχίζεται και θα παρακολουθήσει η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βέμπστερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες. Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Πάμε στο σημείο 7, ετήσια έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τον Απρίλιο άλλαξε ο εσωτερικός κανονισμός του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 54, Επιτροπή ΕΚΟΝ και Επιτροπή Προϋπολογισμών ανέλαβαν την εξουσία να εκπονούν ετήσια έκθεση όσον αφορά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η ΕΚΟΝ και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθεμία με τη σειρά της θα εκπονεί την ετήσια έκθεση. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να παρακολουθεί το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όσοι ταξιδεύατε μέσω αντιπροσωπιών και πήγατε στις χώρες εταίρου, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα γνωρίσετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όλο και περισσότερο γίνεται σημαντική και εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον πραγματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στο νέο πακέτο εξωτερικών επενδύσεων που θα αφορά συνεργασία ιδιωτικού ε, και δημοσίου τομέα. Ο κύριος Λούκε έχει μελετήσει το θέμα, είναι ο συγητής μας και θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν στην προηγούμενη συνεδρίαση που έπρεπε να παρουσιαστεί η έκθεση. Η γνωμοδότηση που, η άποψη που εκφράζει στην έκθεσή μου είναι εν γέννη θετική όσον αφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις συναφείς πολιτικές. Είναι πολύ καλό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο ε, δίνει τις χορηγίες μαζί με τις ε, χορηγίες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι των ετουσομένων χωρών και αυτό εξυπηρετεί το σκοπό της κρίζωσης της ένδυας. Αν θέλουμε να έχουμε σφαιρική ανάπτυξη για όλους, μέσω βελτίωση των υποδομών, στήριξη ιδιωτικού τομέα, μέσω περιφερειακή ολοκληρώσεω και μειώσεω των συνεπειών τη αλλαγή του κλίματο. Τρία βασικά σημεία εμπεριέχονται με επικρίσεις ή συστάσεις. Πρώτον, ο ρόλος των μικρών πιστώσεων, μικροπιστώσεων. Από την έκθεση βλέπουμε ότι οι μικροπιστώσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όσον αφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στηρίζει η θέση απασχόλησης, στηρίζει την απασχόληση των γυναικών και είναι αποτελεσματικότερη μέθοδος από άλλα μέτρα. Οι μικροπιστώσεις όμως είναι μικρό, πολύ μικρό ποσοστό των δανειδοτήσεων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σχετίζονται με τις χώρες ΑΚΕ. Λόγω της επιτυχίας των μικροπιστώσεων, ζητώ διάθεση περισσότερων πόρων για μικροπιστώσεις τις όμενες χώρες και όχι μόνο στις χώρες Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού. Προσμέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων της Ευρωπαϊκής Τάξης Επενδύσεων είναι κάτι καλό, αυξάνει τη διαφάνεια, ο έλεγχος. Όμως το σχετικό πλαίσιο ελέγχου περιορίζεται σε αξιολόγηση και εκτίμηση. Για να αυξηθεί διαφάνεια και ο έλεγχος, ζητώ εκ των υστέρων αξιολόγηση δείγματος έργων που έχουν υλοποιηθεί. Και αυτό να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Αυτή η σύγκριση με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να υποβάλλεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Εξίσου σημαντικό η βελτίωση των πληροφοριών για την εξολόγηση προγραμμάτων. Να μην ευνοούνται οι μεγαλύτερε επιχείρησει εναντίον των μικροτέρων. Να μην αναφέρονται μόνο θέσει απασχόληση που δημιουργούνται και στηρίζονται, αλλά και εκείνων που δημιουργούνται μέσω των διαφόρων προγραμμάτων. Τρίτο σημείο. Η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν αναφέρει δυστυχώς τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας αυτής πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. Πρέπει να υπάρχει μία ετήσια έκθεση περί αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νόρμπερτ πρώτος και μετά η κυρία Χάταλα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του κυρίου Φραντσουλίκα Θέλω να πω το εξή, ότι ενδιαφέρεται πολύ να συνεργαστεί μαζί σα για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθεται την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στι αναπτυσσόμενε χώρε. Η τράπεζα αυτή πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των επιχειρήσεών τη και να εστιαστεί σε ποιοτικά προγράμματα που έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Η τράπεζα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη περιοχής, της περιοχής των χωρών ΑΚΕ Ζητείτε από την τράπεζα να εστιάζει τα στηριότητές της επί στήριξης των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας του ΙΕ. Πρέπει η τράπεζα να προσέξει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις προσπάθειες που καταβάλει και πρέπει να έχει θεμητή διαχείριση των προγραμμάτων. Πρέπει οι πολιτικές της και τα προγράμματά της να ευθυγραμμίζονται με στρατηγικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και το σχέδιο δράσεω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ταιριάζουν τα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να επεκτείνει τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζομένων κοινοτήτων όσον αφορά τι επενδύσει σε φυσικού, φυσικούς πόρους και αιγαίε Το Δεκέμβριο του 2015 εκρήθη μια στρατηγική της Τράπεζας για την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος. Τα προγράμματα για την καταπολέμηση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να είναι στο 35% των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020. Πρέπει να εξασφαλίζει η Τράπεζα ότι τα μέτρα της και τα προγράμματά της πρέπει να βασίσουν σε κριτήρια επιλεξιμότητας για τις δράσεις για το κλίμα και οι πτυχέ του κλίματο πρέπει να ενσωματώνται σε όλε τι προσπάθειες που καταβάλει η Τράπεζα εκτό Ευρώπη. Πρέπει να εξασφαλίζεται επίση ότι οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν επενδύονται σε φορείς τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα διαφάνειας. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να προχωρήσει πιο πέρα όσον αφορά τις ισχύουσες ε, απαιτήσει περί διαφανείας, για να μην υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Πρέπει η τράπεζα να έχει ε, μέχρι το 2017 ένα πρόγραμμα φορολόγησης και να προσέχει όταν συνεργάζεται με διάφορες νομοθεσίες και διάφορες χώρες ότι οι χώρες συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές περί δίκαιης φορολόγησης η Ευχαριστούμε για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που ετοίμασε ο συνάδελφος Λούκε. Πολλά από τα υποθέντα που εξέφρασε ο κ. Φαντσουλίτσα με βρίσκουν σύμφωνοι. Αυτά που διάβασε ο Νόρμπερτ. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Διότι θα παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο, Ευρωπα... στο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων που θα συζητήσουμε και άλλες φορές αυτή την εβδομάδα. Από την πλευρά μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η τράπεζα είναι σε θέση να εφαρμόσει και να χρηματοδοτήσει ποιοτικά προγράμματα που δίνουν πραγματικά αποτελέσματα στον αφορά την ανάπτυξη. Άρα, πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η τράπεζα ήδη εργάστηκε σκληρά όσον αφορά τα μέτρα διαφύλαξης για τα κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θέλαμε να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά. Επίσης, καλό ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ετοιμάζει μια στρατηγική με βάση την ισότητα των φύλων. Ο συνάδελφος Λούκε το ανέφερε αυτό. Ξηρίως μέσω της μικροχρηματοδοτήσεως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προώθησε την απασχόληση των γυναικών. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, ε, διότι στις χώρες στις οποίες κινείται η τράπεζα υπάρχουν προβλήματα ανισότητας ανδρών και γυναικών. η τράπεζα απομακρύνεται από τα ε, ανθρακοβόρα προγράμματα στις χώρες αυτές. Κυρίως όταν έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Συμφωνία των Παρισίων η αλλαγή του κλίματος. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι σοσιαλιστές για τη συνεργασία. με τους σηματοψηφιτικούς μεσάζοντες που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά φορολογική διαφάνεια η συνεργασία σε φοροδιαφυγή και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Και ελπίζω ότι η γνωμοδότησή μας θα οδηγήσει σε ενδελεχέστερες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Μπορούμε να καλέσουμε μέλη της Επιτροπής να έρθουν να μας εξηγήσουν. Αν μιλήσω πιο δυνατά, αν ουρλιάξω θα με ακούσετε. Δεν ξέρω αν οι διερμηνείς μ' ακούνε καθαρά, όχι. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, να αυξήσουν το, την ένταση των μικροφώνων. Τώρα που ήμουνα, μπερδεύτηκα. Μπορούμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έρθει. Πράγματι αλλάζει ο ρόλος τη σε σχέση με το παρελθόν και αρκετά. Στα άτυπα συμβούλια συμμετέχουν τακτικά διότι είναι αναμειγμένη στο εξωτερικό σχέδιο δράση η τράπεζα αυτή. Ελπίζω να αναλύσουμε ει βάθο το νέο σχέδιο, το φθινόπωρο. Χρειάζονται περισσότερε επαφέ με την τράπεζα. Δεν έχω άλλου ομιλητέ. Α, καλύτερα. Δυνάμωσε ήχο. Ευχαριστούμε τους τεχνικού. Κύριο Σιάφος, από τη Γενική Διεύθυνση, κύριος Κράβος, Σιάφος από την ΤΕΦΚΟ και κάποιος ανώνυμος από την ε, Οικονομική Διεύθυνση. Ο κ. Σιάβος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για την έκθεσή τους. Αυτό είναι ένα θέμα βεβαίως που αφορά κυρίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εδώ δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε αυτό το οποίο αναφέρει η έκθεση, ιδιαιτέρως όσον αφορά την έμφαση που δίδεται, που θα πρέπει να δοθεί, ούτε ώστε να εξασφαλίσουμε ε, μια πιο αποτελεσματική εργασία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης ούτω ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την εξάλληψη και την ελάφρυνση της, ανακούφιση της φτώχειας. όσο δυνατόν, σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα εδώ. Και βεβαίω ο σημαντικός ρόλος θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επενδύσεων θα συζητηθεί σε μια ειδική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Δεν έχω το όνομά σα ίσως να μας συστηθείτε. Λέγομαι Μετέο Ρίτσο, είναι από το ΕΚΟΦΙΤ και θα ήθελα ε, να πω ότι συμφωνώ με τον ε, προλαλήσαντα. Χάιντι, βεβαίως θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν είχαμε τις απαντήσεις σε κάποιες από ερωτήσεις που θέσαμε. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων εδώ όσον αφορά τη χρήση αυτών των πιστώσεων και ίσως ε, θα μπορούσατε να σχολιάσετε εδώ για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά την ασφάλεια. Ναι, απάντηση. Οι χώρες ε, πιέζουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μειώσουν ε, την ε, δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν χαμηλότερη φορολόγηση. Και ίσως θα, ήταν, θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις μετά την συζήτηση που θα γίνει με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά κατά πάσα πιθανότητα μετά θα είμαστε σε θέση, μετά από αυτή τη συζήτηση ε, ναι, αλλά όσον αφορά την ε, πολιτική για τα εχέγγυα, για τις δικλείδες ασφαλείας, απάντηση. Ε, πιστεύω ότι δεν είμαι το ενδεδειγμένο πρόσωπο να απαντήσει. Νομίζω ότι όποτε συζητούμε αυτό το ε, πρόγραμμα, το εξωτερικό επενδυτικό πρόγραμμα, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα, αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι σημαντικά. Ε, κύριε Λούκια, έχετε κάτι να προσθέσετε? Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δώσω την προσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Είναι η 11η Οκτωβρίου, αύριο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου στην Επιτροπή. Ε, δεν ξέρω αν θα φτά, μας φτάσει ο χρόνος είναι κάπως στενά τα περιθώρια. Αύριο λοιπόν στις 12 θα πρέπει να κατευθούν οι τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούκε. Ολοκληρώνεται εδώ η, η συζήτηση. Και, εδώ το... και τώρα έχουμε το επόμενο θέμα, την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε μια προσκεκλημένη ομιλήτρια, ε, αλλά νομίζω ότι δεν παρευρίσκεται εδώ, γι' αυτό θα πρέπει να διακόψουμε τις εργασίες μας για μισή ώρα. Βεβαίως είναι κάπως ε, ενοχλητικό αυτό, αλλά παρόλα αυτά έως παρατέταρτο εάς διακόψουμε.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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

να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

Okay, colleagues, we're going to because it's, we said we start at quarter and um, we need to stick to our... Ε, συνεχίσουμε γιατί είναι παρατέταρτο και να μην ε, χάνουμε χρόνο. Ε, σημείο 8 τώρα, πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και πώς διασφαλίζουμε την πρόσβαση στην ε, προσιτή κατάλληλη ενέργεια. ένας από τους ε, βασικούς ε, στόχους ε, του έβδομου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω και τότε ο Επίτροπος είχε τότε θέσει αυτό το ζήτημα, το έχει αρχίσει ως σημαντική προτεραιότητα στο συνολικό πρόγραμμα. Βλέπετε ότι πολλές φορές θέτουμε τέτοια ζητήματα, πρόσβαση στην ενέργεια και ο Νόρμπερτ στο παρελθόν το έχει εξετάσει. Οι συντονιστέ λοιπόν συμφώνησαν να ε, συντάξουμε ένα προφορικό ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσουμε ακριβώ τι συμβαίνει ω προ την πρόσβαση στην ενέργεια. Γιατί δεν έχει νόημα να το έχουμε ω προτεραιότητα για τρία-τέσσερα χρόνια και μετά να το ξεχνάμε γιατί ε, ανακύπτουν νέε προτεραιότητε. Γιατί η πρόσβαση στην ενέργεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Πριν εγκρίνουμε όμω την προφορική μας ερώτηση που θα τεθεί στην επόμενη συνεδρίασή μα, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο σε έναν εμπειρογνώμονα για την πρόσβαση στην ενέργεια. Έχουμε καλέσει την Molly Haley από την Smart Villages. Θα εξηγήσω ακριβώς τη Molly να μας εξηγήσει τι είναι αυτά τα έξυπνα χωριά προσπαθούν ουσιαστικά να έχουν ε, ε, κατάλληλη τεχνολογικά ενέργεια στα, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσουμε το λόγο στη συνέχεια. Παρακαλώ, μόλι έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την πρόσβαση στην ενέργεια και τις ευκαιρίες και προκλήσεις σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του 7ου στόχου από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Smart Villages είναι μια ε, πρωτοβουλία τριών ετών που θέτει ότι ε, ακόμα και τα απόμακρα σημεία μπορεί να είναι πολύ καλά σημεία να ζει κανεί ε, με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην ενέργεια, ε, δυνατότητε απασχόληση για άντρε και γυναίκε ε, και ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Και εμεί θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι ένα φορέα διευκόλυνση τη ανάπτυξη και στο πλαίσιο των στόχων αναβιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ε, μετάβαση και αστιφιλία. Όμως ε, θεωρούμε ότι ε, έχουμε ακόμα περισσότερε ευκαιρίες να διερευνήσουμε από την πρόσβαση στην ενέργεια αλλά και με μια διακλαδική προσέγγιση. Η πρωτοβουλία μας έχει διοργανώσει 25 εργαστήρια με πάνω από 500 φορείς του κλάδου, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επιστήμονες, ερευνητέ. Ε, και επιχειρηματίες για να κατανοήσουμε και τις προκλήσεις για ε, τα ε, έξυπνα χωριά αλλά για να δούμε και ποιες μπορούν να είναι λύσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με τα εθνικά και περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα. Ελαμβάνουμε χρηματοδότηση από δύο ιδρύματα και στο Cambridge και στι ΗΠΑ. Είναι πολύ καλό που έχουμε αυτόν τον 7ο στόχο ε, βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και άλλου διασυνδεμένου ε, στόχου. Όμω, μία από τι προκλήσει είναι αυτού του 7ου στόχου είναι ότι δεν ορίζει το ελάχιστο επίπεδο ε, οικουμενικής πρόσβασης στην ενέργεια. Θα είναι μια μινιμαλιστική προσέγγιση ή πιο φιλόδοξη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, επιλέξουμε το ελαχιστο επιπεδο οικουμενικη πρόσβαση στην ενεργεια και πιο φιλοδοξη Εμεί πιστευουμε οτι πρεπει να ωφελεί αυτούς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ωφελει αυτού που διατρεχουν μεγαλυτερο πίσω. Ε, και σε ε, που χρειάζονται αυτές τις αποκεντρωμένες λύσεις, γιατί το δίκτυο δεν θα τους ε, καλύψει για πολλά χρόνια. Τι εννοούμε με ε, φιλοδοξία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ συνάντησα τον Μάρτιν Κυριόγκη το 2014 στην Ταζανία. Ο Μάρτιν είχε ε, μεγαλώσει στις παιδιάδες της Τανζανίας, μετά σπούδασε στο Δουβλίνο και στο Ινωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του ήθελε να ξεκινήσει έναν ε, ραδιοφωνικό σταθμό για να ενημερώνει τους Μασάι για ε, την κατάστασή τους και για την προστασία των γεών τους. Όμως για να το κάνει αυτό χρειαζόταν ενέργεια. Όμως πέραν του ραδιοφωνικού σταθμού ε, είδε ότι οι νέοι και οι νέε συνεχώς κατευθύνονταν προς τις πόλεις και δεν υπήρχαν αρκετές λύσεις για απασχόληση. Πήγε ξανά λοιπόν στην Τανζανία σε ένα χωριό που λέγεται Τέραντ που τότε ήταν μια τελείως απομακρυσμένη περιοχή χωρίς ε, τρεχούμενο νερό και ρεύμα. Και ο κόσμος πραγματικά πίστευε ότι ήταν τρελός. Όμως είδε την ε, ευκαιρία να σταματήσει αυτή τη ε, μετατόπιση των Μασάι προς τις πόλεις και να τους βρει και δουλειά. Ε, ίδρυσε λοιπόν μία οργάνωση, την IOPA, ε, και χάρη σε φιλανθρωπία από συγκεκριμένους οργανισμούς στην Ολλανδία, από, από ένα, μια γεννήτρια 40 κιλοβάτ, ε, κατάφερε να φτιάξει μια ολόκληρη μονάδα παραγωγής, ενέργειας, αλλά και έναν διαφωνικό σταθμό, ε, αλλά και μονάδα παραγωγής ε, τυριού, γιαουρτιού, με πολλές μικρές επιχειρήσεις, κομμωτήρια, και έδινε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε καλύτερη παιδεία. Όπως και με άλλα μικροδίκτυα βέβαια, παίρνει χρόνο η όλη διαδικασία επιστροφής ε, της επένδυσης ε, των χρηματοδοτών. Όμως θεωρήσαμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και ακόμα και τους επενδυτές τελικά θεωρήθηκε καλό, γιατί ας πούμε οι τεροπαραγωγοί έχουν ε, λάβει ε, πολλά βραβεία για τα προϊόντα τους. Το τέρατ λοιπόν έχει ενισχυθεί με όλη αυτή τη διαδικασία. Περίπου μισή από τους ε, νέους που έφευγαν για τις πόλεις είτε δεν έφευγαν πλέον ή και επέστρεφαν στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου και οι γυναίκες διαδραμάτιζαν πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία και στη φιλοσοφία του προγράμματος. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η ενέργεια αυτή ε, αξιοποιείται για παραγωγικούς σκοπούς. Δηλαδή θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές και το εισόδημα των κατοίκων και έτσι γίνεται βιώσιμο και ένα χωριό. Μεγάλη έμφαση δίνεται στους νέους και στις γυναίκες στην προσέγγιση τους. Το τέρατ είναι λοιπόν ένα υπόδειγμα εναλλακτική όπου έχουν την επιλογή οι κάτοικοι να μείνουν ε, στο χωριό τους ή να πάνε στην πρωτεύουσα καθώς το επιθυμούν. Εμείς ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους προγράμματα και θα ήθελα στην συντομία να αναγνωρίσω και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν συγκεκριμένε επιχειρήσεις, ε, οργανισμοί. Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα όλων αυτών που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο και θα ήθελα να κάνω μια μικρή μνήα στο έργο τους. Παρότι δεν μπορώ να επισέλθω τις λεπτομέρειες, ή ίσως μπορούμε να το αναλύσουμε περαιτέρω στη συζήτηση. Σίγουρα γνωρίζετε πολλές αυτές τις εταιρείε και οργανισμούς ε, που μπορεί να ασχολούνται με την ηλιακή ενέργεια, ε, την κινητή τηλεφωνία, ε, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις καθαρές τις οικολογικές δηλαδή, ε, ή άλλες που ασχολούνται με μικροδίκτυα, με ηλιακές αντλίες, αλλά και την ε, αιωλική αλλά και την ενέργεια. Αναγνωρίζουμε τρόπους με, τον, με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών έχουν συμβάλει σε αυτό το εγχείρημα μέσω της παραδοσιακής αναπτυξιακής ε, χρηματοδότησης ή με άλλες πιο δημιουργικές μεθόδους, με μερική χρηματοδότηση για παράδειγμα. κάτι τώρα που ε, έχει προκύψει ε, πρόσφατα είναι μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία ε, που πραγματικά θεωρούμε πολύ θετική για το μέλλον και είναι λίγο πιο φιλόδοξη και νομίζουμε ότι και ο Επίτροπος Επίπορξ αυτό είχε κατά νου όταν αναφερόταν σε αυτό το ζήτημα. Και βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν εύκολη οδός και για τους ε, χορηγούς, γιατί τα προγράμματα δεν είναι πάντα επιτυχή. Όμως αυτό δεν είναι κακό, γιατί μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας. Αντί να, μείνω, εδώ, θα ήθελα ε, να σας ε, αναφέρω ορισμένα στοιχεία που ε, μας βοηθούν στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια είναι σε επίπεδα επαρκή για την αξιοποίηση αυτών των παραγωγικών σκοπών και αυξάνει τα εισοδήματα. Για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα ε, ενέργειας είναι πραγματικά αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα σε αυτές τις ε, κοινότητε. Βέβαια, πρέπει να λύσουμε το θέμα της χρηματοδότησης και για τους επιχειρηματίες. Όπως ξέρετε, χρειάζεται ε, κεφάλαιο για να γίνουν αυτά τα προγράμματα πρέπει να διασφαλίσουν κεφάλαιο και άλλε ε, μορφές χρηματοδότησης και δανειοδότηση, γιατί δεν παίρνουν δάνεια από τράπεζε συνήθω. Αλλά και με τοπικέ ε, τράπεζε θα πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε ακούσει από πολλού ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα οικοδόμηση δυναμικού ε, μεταξύ των τοπικών αρχών. Πολλοί απλώ δεν κατανοούν τον δμό ε, τον κλάδο μάλλον, τον off-grid, ενεργειακό κλάδο εκτό δικτύου. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι χρειάζονται και άλλες ε, δημιουργικές μορφές. και ότι αυτά τα, ακόμα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα φτάνουν τις πλέον απομακρυσμένες ε, περιοχές και προγράμματα. Ξέρουμε ότι στην Ανατολική Αφρική Μία από τις πλέον αναπτυγμένες ε, ε, αγορές είναι αυτή για την ε, οικιακή ηλιακή ενέργεια. Όμως δεν έχει επεκταθεί το πρόγραμμα όσο θα θέλαμε και εκεί και σε άλλες περιοχές. Ξέρουμε επίσης ότι τα έξοδα συναλλαγών είναι πάντα πολύ υψηλά, καθώς και η επεξεργασία αυτών των προγραμμάτων. Θέλουμε να βρούμε ε, τρόπο καλύτερης κατανομής ε, των ε, πόρων. Ένας επιχειρηματίας που ξέρω εγώ και ασχολείται ακριβώς με την εκτός δικτύου ενέργεια για την επεξεργασία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ανέφερε πρόσφατα την ιδέα ε, στενότερης συνεργασίας με τους λεγόμενους angel investors. Ε, βλέπουμε ότι αυτοί που επενδύουν ε, έχουν και άλλα κίνητρα εκτός από την επίτευξη κερδών και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο εδώ. Στις κυβερνήσεις βλέπουμε επίση την ανάγκη οικοδόμησης δυναμικού για να βελτιώσουμε την κατανόηση των ωφελών αλλά και την ε, ενθάρρυνση των ενεργειακών επιχειρηματών, για παράδειγμα. Η επιχειρηματικότητα δεν ενθαρρύνεται και δεν στηρίζεται πάντα από τι εθνικέ κυβερνήσει. Πρέπει να βρούμε τρόπου να το αλλάξουμε αυτό. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι για να πετύχουμε το στόχο μας χρειαζόμαστε και καθοδήγηση και από ε, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πρέπει να σταματήσουν οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε δύο επίπεδα επιχειρηματικότητα εδώ. Οι ε, επιχειρηματίες ενέργεια, στον κλάδο της ενέργειας που ε, φτάνουν και φέρνουν αυτά τα προγράμματα στα χωριά, αλλά και σε αυτά τα χωριά μέσα υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες που, με μικρές επιχειρήσεις που μπορούν όμως να δώσουν μια νέα όθηση ε, σε αυτό το στόχο. Και νέες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ιδρυθούν. Χρειαζόμαστε ε, συμμετοχή και οικοδόμηση εμπιστοσύνης για πρωτοβουλίες από τα κάτω προς τα πάνω ε, και πρέπει, αυτό είναι απαραίτητη προπόθεση για να έχουμε βιώσιμα προγράμματα. Και από οικονομική πλευρά, για του καταναλωτέ, για του κατοίκου αυτά τα χωριά, κάποιε φορέ ε, είναι δύσκολο να κρίνουμε τι μπορεί κανείς ε, να πληρώσει. Τι είναι προστό δηλαδή για τον ε, καταναλωτή. Κάποια συστήματα έχουν... Κάποια προγράμματα έχουν συστήματα με βάση την κατανάλωση, όμως αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Γι' αυτό κάποιες φορές ε, βλέπουμε κοινότητες που θέλουν να αγοράσουν γεωργικά μηχανήματα για να αξιοποιήσουν αυτή την ενέργεια για να έχουν για παράδειγμα ένα μήλο ή να ε, ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία παραγωγής. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτοί που ενδέχεται να γίνουν μικροεπιχειρηματίες δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν τα υψηλά επιτόκια. Χρειάζονται προσβάσιμα, προσιτά επιτόκια για να μπορούν να τα επεξέλθουν. Σε ό,τι αφορά τεχνολογία τώρα, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη προ την τεχνολογία βέβαια. Κάποιοι στο παρελθόν είχαν αρνητικέ εμπειρίε με χαμηλή ποιότητα προϊόντα ή ακόμα και πλαστά ε, ή μη ποιοτικά τέτοια προϊόντα. Αυτό είναι σημαντικό ε, για τους υπεύθυνου χαράξης πολιτική και τι ρυθμιστικέ αρχέ αυτών των χωρών. Κάποιε φορές δεν είχαν ε, τεχνική υποστήριξη και αυτό είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο. Όμω πρέπει και οι ίδιοι ε, να καταρτιστούν για να διατηρήσουν τεχνολογία Ε, κάποιες φορές υπάρχουν και γραμμές τεχνικής υποστήριξης και άλλα εργαλεία. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτό που χρειάζονται, το που χρειάζεται οποιοδήποτε έχει ένα τεχνολογικό προϊόν, είναι και τα ανταλλακτικά, για να μπορούν να, να διορθώσουν ένα πρόβλημα. Γι' αυτό ορισμένα προγράμματα έχουν ε, αποτύχει και είναι εύκολο να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα. Τέλο, οι επιχειρηματίε του χωριού χρειάζονται την οικοδόμηση δυναμικού και για τα δικά του επιχειρηματικά σχέδια. Χρειάζονται λοιπόν ε, ε, συμβουλευτική και καθοδήγηση για το πώ θα φτιάξουν τι επιχειρήσει του, να βρουν τι καλύτερε μορφέ ε, εισοδήματο και να έχουν πρόσβαση σε αγορέ. Κλείνοντα. Το πιο σημαντικό είναι πώ θα συνεργαστούμε με του επιχειρηματίε να λύσουμε το θέμα τη χρηματοδότηση, ώστε οι χωρικοί να έχουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματο η οικοδόμηση δυναμικού είναι κρίσιμη σημασία για όλου του εμπλεκόμενου. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε θα πρέπει να συνδέονται και με πρωτοβουλίε στι υπηρεσίε. Υγεία, εκπαίδευση, καθαρό νερό και ε, παραγωγική σκοπή για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη τα αναπτυξιακά. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο δρόμος. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ και ε, περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα κάνουμε και αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα των έξυπνων χωριών έχω αφήσει ορισμένα φυλάδια στη γραμματεία τα οποία μπορείτε να δείτε μπορώ να σας στείλω και μέσω mail αν ενδιαφέρεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα ζωντανά παραδείγματα που μας δώσατε όσον αφορά το τι συμβαίνει με διάφορα προγράμματα. Μοιραστήκαν τα φυλάδια στους συναδέλφους. Πρέπει να σας έδωσε ο αρμόδιος υπάλληλος ε, το φυλάδιο. Νόρμπερτ Νόισερ. Α, Πολ Ρούμπικ πρώτος και μετά ο Νόρμπερτ Νόισερ. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί πιστεύω ότι αυτή η ομιλία για τα Smart Villages ακριβώς μας ε, έδειξε προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Και νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν εδώ για όλους μας έχουν τεράστια σημασία ε, γιατί πραγματικά έχουν επιλεγεί σωστά οι προτεραιότητες. Βεβαίως χωρίς, την, ε, χωρίς ενέργεια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη. Χρειάζεται η ενέργεια για τις τηλεπικοινωνίες, χρειάζεται ενέργεια για τον ε, τομέα της υγιεινής και για την ασφάλεια των γυναικών χρειάζεται ενέργεια. Ε, αν δεχτούμε ότι υπάρχουν χώρες όπου είναι νύχτα 12 ώρες, βλέπουμε πόσο απαραίτητη είναι η ενέργεια. Άρα η ενέργεια είναι η βάση ε, μπορεί να, σχέση με την οποία μπορεί να προσμετρηθεί η ευημερία. Χρειάζεται λοιπόν ενέργεια κυρίως στην ύπεθρο και στα μικρά χωριά και στις περιφέρειες γιατί ε, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξουν περιφερειακές υποδομές και αποκεντρωμένες δομές όπως είναι ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια κλπ. Ε, projects τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε επίπεδο κοινοτήτων. Χρειάζονται λοιπόν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που μπορούν να παράσχουν κάποια κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις. Και βεβαίως όπως έλεγχε είναι σημαντικό να ρυθμιστεί και το ζήτημα του σέρβις αυτών των εγκαταστάσεων γιατί μόνο με τις ε, καθαρές επενδύσεις γρήγορα οι εγκαταστάσεις τελματώνουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν κάποια μοντέλα τα οποία να περιλαμβάνουν και το σέρβις αυτών των εγκαταστάσεων. Και εδώ είναι χρήσιμο να δούμε τις μικρές οικογενειακές ε, μονάδες, έτσι όπως τις δείξατε στα διαφάνειές σας να δημιουργηθούν λοιπόν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, τέτοιου είδου μοντέλα. Και ε, βεβαίως να, να γίνονται ε, με διαφάνεια οι προκηρύξεις διαγωνισμών, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν μικρές επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε ότι οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι ε, συχνά στις πόλεις μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, αλλά δεν ενδιαφέρονται για πιο μικρές δομές. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι δικό μας μέλημα να προθίσουμε ακριβώς τις ε, μικρές αυτές δομές, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, ε, ανθρώπους δηλαδή που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ήδη ίδιοι την εκπαίδευσή τους και την επαγγελματική κατάρτιση και να τεθεί αυτή στο επίκεντρο της προσοχής τους. Ε, και βεβαίως μπορούν να αναζητηθούν και διεθνείς εταίροι όπως είναι η UNICEF για παράδειγμα ή ε, ο διτός τρόπος εκπαίδευσης ο οποίο να συμπεριλαμβάνει ακριβώς ε, και το στοιχείο αυτό της, ε, του σέρβις, όπως σας είπα, την, των εγκαταστάσεων. Ευχαριστούμε. Νόρμπερτ Νόισερ. Ευχαριστούμε και πάλι για την, ε, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και φαντάζομαι και έγινε αισθητό, αισθητός ο, ο με τον οποίο προσεγγίσετε αυτή τη θεματολογία και μπορεί πραγματικά να προωθήσει την αναπτυξιακή συνεργασία. Το 2012 Υπήρξε μια έκθεση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η βασική στόχη τότε ήταν να επικεντρωθούμε με την ευρωπαϊκή μας πολιτική σε μικρές ε, περιφερειακές ε, και ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Όπως είπε ο συνάδελφος, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, συγκεντρώνονται στις ε, αστικές περιοχές και στις πόλεις, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στις περιοχές της Επέθρου που δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στην ενέργεια. Μία επιτυχής πολιτική στον τομέα αυτό θα σήμαινε και μία αναστροφή της τάσης της αστικοποίησης. Γιατί ε, βλέπουμε πως τα μεγάλα κεφάλαια μεγεθύνονται συνεχώς. Αν δούμε τι γίνεται στο Λάγος ή στην Κινσάσα, όπου όλοι οι άνθρωποι πάνε στις ε, πόλεις, όπου έχουν μια καλύτερη προοπτική. Με την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενέργεια θα μπορούσαμε να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση και ίσως και να την αναστρέψουμε σε ορισμένους τομείς. Σημαντικό εδώ είναι ότι η ενέργεια είναι βιώσιμη, όπως είπαμε, και η Αφρική ιδιαίτερως αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ε, προσφέρουν εδώ όσον αφορά την ε, ηλιακή ενέργεια, την αιωλική ενέργεια, αλλά και τα συστήματα υδροδότησης καλύτερες ευκαιρίες από ό,τι στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτές οι ενεργειακές ε, πηγές. Όσον αφορά τους αναπτυσσόμενους στόχους της χιλιατηρίδα, η πρόσβαση στην ενέργεια δεν αποτέλεσε θέμα αλλά εδώ στους διάσημους αναπτυξιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στην ενέργεια και ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε ε, σε ένα άλλο σημείο της ημέρας τη διάταξης να δούμε πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα μέσα των οποίων μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι με μια ε, ενεργειακή εξασφάλιση της ενέργειας μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά στις περιοχές της υπαίθρου γιατί μπορεί να λειτουργήσει ούτε σχολείο ούτε κέντρο υγείας χωρίς ενέργεια ε, το βράδυ μετά τις 6 στην Αφρική ε, πολλές ε, επιχειρήσεις δεν λειτουργούν και λέω 6 γιατί τότε νυχτώνει στην Αφρική. Θα ήταν λοιπόν τεράστιο πλεονέκτημα και για τις γυναίκες όπου θα βεβαίως θα εξασφαλιζόταν ένα καλύτερο επίπεδο προστασία των γυναικών εφόσον υπήρχε φως. Ε, διεθνώς λοιπόν υπάρχει ένα καλό πλαίσιο, Ban Ki-moon με τη δική του πρωτοβουλία Energy for All ε, μέχρι το 2030 ε, διατύπωσε ακριβώς το πλαίσιο της προποθέσεις και τώρα να σε εμά να χαράξουμε από κοινού με την Κομισιόν μια στρατηγική η οποία να εφαρμόζει αυτά τα οποία πέτυχε ο Πίμπαλ στα τελευταία δέκα χρόνια. Και ως Επιτροπή εδώ θα πρέπει να τεκμηριώσουμε ε, την εξέλιξη, τι είδους πρόοδοι σημειώθηκαν μέσα των πρωτοβουλειών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο έζησα εγώ ίδιο. Πήγαμε σε δύο μικρά χωριά στην Κένια και τα δύο αυτά χωριά είχαν περίπου και τα δύο χίλιους ε, κατοίκους και τα δύο είχαν πρόσβαση στην ενέργεια μέσω ε, μιας υδροτουρμπίνας ε, και στα ένα χωριό ε, πραγματικά ήταν ευγνώμονες που είχαν αυτή την πηγή ενέργειας και ε, ρώτησαν τη ΜΚΟ κατά πόσα έχουν λεφτά να φτιάξουν και μια δεύτερη εγκατάσταση. Στο άλλο χωριό οι άνθρωποι εκεί είπαν ότι θέλουμε και εμείς ε, να συμβάλλουμε με χρήματα ε, για το γεγονός ότι μας χαρίσατε αυτή την εγκατάσταση και να αγοράσουμε μόνοι μας μία δεύτερη. Ε, και βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πόσο σημαντική είναι και μία εξαρτή ενημέρωσης για τους κατοίκους. Και εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερος ζήλος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Θεοχάρους, Ελένη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, βεβαίως για μας τους Ευρωπαίους, θα έλεγα στον κύριο Νόιζερ, δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό, εντυπωσιακή εμπειρία από το να βλέπει κανείς τον ουρανό σε μια αφρικανική περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό τριγύρω όπου ανοιχνεύει και το Σαυρό του Νότου και όλους τους αστερισμούς και νομίζει ότι αν απλώσει τα χέρια του θα τριγύσει όλα τα αστέρια του ουρανού. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή δεν είναι η πραγματικότητα για τους ντόπιου κατοίκου εκεί πέρα. Θέλω να συγχαρώ την ομιλήτρια για την επαναστατική ιδέα που έχει εισαγάγει καθώς επίσης και για μια ανάλογη ιδέα που έχει να κάνει με τα περίπτερα, τα ενεργειακά περίπτερα τα οποία εγκαθίστανται βασικά στο κέντρο των μικρών χωριών που δεν έχουν ηλεκτρισμό. Ε, τώρα τελευταία εργάζομαι πάνω σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Ρουάντα για την κατασκευή αυτών των μικρών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας και τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας όχι κατευθείαν σε ηλεκτρισμό αλλά σε θερμική ενέργεια με τη χρήση κατόπτρων και γραφίτη που έχει ως αποτέλεσμα να δουλεύουν τα συστήματα 24 ε, ώρες το 24 ώρο και όχι μόνο τις ώρες που έχει ηλιοφάνεια. Αυτά τα projects χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 10 εκατομμύρια δολάρια και ε, ευρώ και η πρόθεση είναι να εγκατασταθούν τέτοια 10 πιλωτικά προγράμματα σε όλη την Αφρικανική ε, Ήπειρο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που μας παρεμποδίζουν να αντιμετωπίσουμε, να επιτύχουμε το ε, Sustainable Development Goal No. 7. Τώρα, Εκείνο που έχει σημασία όσον αφορά την παροχή ενέργειας στις, ε, αγρο... στις απομακρυσμένες περιοχές είναι ότι το υδροηλεκτρικό δυναμικό της Αφρικής δεν έχει αξιοποιηθεί παρά μόνο στο 5%. Δηλαδή σκεφτείτε τι θα μπορούσε να επιτύχει ο αφρικανικός πληθυσμός αν είχε αξιοποιήσει μόνο την υδροηλεκτρική ενέργεια που μόνο το 5% χρησιμοποιείται πέρα από την ηλιακή, πέρα από την αιωλική, πέρα από όλες τις άλλες σύγχρονες ε, μορφές ενέργειας. Ε, νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τροφοδοτηθεί η αγροτική περιοχή της Αφρικής, οι απομακρυσμένες περιοχές με ηλεκτρισμό, πρώτα πρώτα για να δουλεύουν οι αντλίες. Οι αντλίες άντλησης νερού για τις ε, διάφορες φοιτίες που μπορούν να κατασκευαστούν, για την εκπαίδευση, για τη χρήση του διαδικτύου, για τις επικοινωνίες, για τα μικρά νοσοκομεία της Υπέθρου. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο με γεννήτριες και τις πιο πολλές φορές την πιο κρίσιμη στιγμή μιας επέμβασης διακόπτει την παροχή σταματά να δουλεύει η γεννήτρια και καταλαβαίνετε τι υφίσταται ένας γιατρός εκείνη την ώρα. Επίσης, όλες αυτές οι χώρε και είναι σε αυτό το σημείο που και πάλι θα επανέλθω στην επιμονή μου ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις είναι τόσο διεφθαρμένες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των περιφερειών, δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει ένα ορφανοτροφείο και ένα ε, σχολείο γιατί δεν έχει αυτά τα βασικά στοιχειώδη πράγματα όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμό και νερό. Αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να τροφοδοτήσει ούτε το ορφανοτροφείο ούτε το σχολείο με ηλεκτρική ενέργεια απομένει σε εμά να ξεκινήσουμε από το βασικό, την λειτουργία αυτών των μηχανισμών που πολύ σωστά έχετε περιγράψει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πείνα, την υποανάπτυξη και να δώσουμε στους κατοίκους καθαρό νερό, συνθήκες υγιεινής, τρόφιμα, εκπαίδευση κυρίως και νοσοκομιακή περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την καλή ομιλία. Νομίζω ότι με το Smart Villages πραγματικά ε, μπορέσατε να εκφράσετε αυτό το οποίο, ε, στο οποίο αποσκοπούμε στην ύπεθρο ε, της Αφρικής, δηλαδή μία αποκεντρωμένη παροχή ενέργειας μέσω μικρών δικτύων στην ύπεθρο. Ε, και νομίζω ότι πραγματικά όλοι οι ομιλητέ ε, αναφέρθηκαν ε, στη βαρύτητα αυτού του θέματος και θα πρέπει και εμείς να υποστηρίξουμε αυτά τα projects ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενέργεια σε αυτές τις περιοχές. Στο Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφιστεί και ένα ψήφισμα το οποίο το σχέδιο ήδη υπάρχει και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή βάση. Αλλά να αποβλέπουμε εκεί σε αυτά τα οποία αναφέραμε σήμερα εδώ, σε μικρέ δομέ ενέργεια, νομίζω πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στην έκθεση αυτή. Γιατί όταν αναφέρεται εκεί μόνο ε, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, δεν εξεδικεύεται η μορφή ότι θέλουμε ακριβώ αυτέ τι μικρέ ε, δομέ. Ε, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, αιωλική ενέργεια κλπ. κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να το διατυπώσουμε συγκεκριμένα. Ε, όλοι ξέρουμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ε, διώχτηκαν από τις περιοχές τους για να κατασκευαστούν ε, φράγματα για παράδειγμα και τις ιστορίες δεν θέλουμε να ακούσουμε στο μέλλον. Το 2000, ε, στις 16 Νοεμβρίου του 2000 ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μία έκθεση, ένα νέο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα φράγματα ακριβώς. Γνωρίζουμε λοιπόν ε, ποια είναι τα προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει, εάν αποβλέπουμε σε αυτές τις μικρές δομές, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για δομές μικρής κλίμακας, small scale. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, πτυχές και να προσμετρηθούν οι δυνητικοί ε, κίνδυνοι. Ε, για παράδειγμα, όταν ε, κάποιοι χωρικοί, κάποιοι αγρότες λιμοκτονούν γιατί καλλιεργούν στα χωράφια τους μονοκαλλιέργειες που προορίζονται για την εξαγωγή. Επίσης η οδηγία για τις ανώσιμες ε, πηγές ε, ενέργειας και εδώ υπάρχουν ελλείμματα και χρειάζονται, ε, υπάρχει μια ανάγκη αναθεώρηση όσον αφορά τη βιομάζα. Νομίζω ότι το ζήτημα του άνθρακα είναι ένα τεράστιο ζήτημα στην Αφρική γιατί δημιουργούνται πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα και αν θέλουμε να τα προβλάβουμε ε, θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια εναλλακτική επένδυση σε μικρές ε, δομές όπου οι αγρότες θα καλύπτονται χωρίς να, είναι, να χρειάζεται να αποψηλώνουν τα δάση για να χρησιμοποιήσουν την ξυλία. Τώρα, όταν έχουμε επενδυτές υπάρχουν ζητήματα κακοδιαχείρισης και εσφαλμένων επενδύσεων ε, το κέρδος ε, είναι ένα ζήτημα εδώ και αυτό θα πρέπει να το δούμε γιατί στα μικρά προγράμματα δεν υπάρχει τέτοιος ε, δεν εξασφαλίζεται συχνά αυτό το κέρδος. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε τα μικρά project ε, θα πρέπει πράγματι να τα κατονομάσουμε έτσι στην έκθεσή μας. Όσον αφορά την εξασφάλιση της οικουμενικής ε, πρόσβασης στην ενέργεια, θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή, από τα, να φύγουμε από τα μεγάλα προγράμματα προς ε, αποκεντρωμένες ε, μικρής κλίμακας λύσεις και δεν θα πρέπει ούτε άμεσα ούτε έμεσα να προωθήσουμε ε, την πυρηνική ενέργεια και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει ξεκάθαρα να ονοματιστεί στην έκθεση και στην περίπτωση αυτή θα έχουμε μια καλή βάση για αυτά τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε ακριβώς στον τομέα αυτό. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα. Ο κύριος Φελίτσε Τσακέο θα πει κάτι. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τα μικρότερα προγράμματα. Ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε εν συντομία τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια ερώτηση. Ξέρω ότι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ μέσω της DG Clean ένα δίκτυο πόλεων σε σχέση με την ενέργεια. Υπάρχει κάτι για χωριά. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η Μόλη δεν πήρα το λόγο πριν. Όταν αναφέρθηκε στην ηλεκτροδότηση ήταν το τελευταίο παράδειγμα του τεράστιου έργου που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη βιώσιμη ενέργεια και την πρόσβαση σε αυτή. Είπατε ότι ο Επίτροπος κ. Πίμπας είχε αναλάβει υποχρεώσεις για την αλλαγή, το θεματολόγιο αλλαγή και θέσαμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ενέργεια για ανάπτυξη βιώσιμη και δημιουργή θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστατούσε στις προσπάθειες της πρωτοβουλίας για βιώσιμη ενέργεια. Ανέλαβε υποχρέωση να υποστηρίξει την σφαιρική πρόσβαση, γενική πρόσβαση στον πληθυσμό μέχρι το 2030 και καταπολέμηση τώρα της αλλαγής του κλίματος και οι πρόσφατες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν στην προτεραιότητα, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ακούσαμε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Πρωτοβουλίες εκτός δικτύου για τα χωριά, το off-grid, για τα χωριά. Ποια είναι η επιτόπια κατάσταση. ακούσαμε και τη σημασία που έχει να αισθάνονται οι χώρες ότι ιδιοποιούνται την πρωτοβουλία αυτή να δημιουργούν ε, κίνητρα για επενδύσεις κάθε κλίμακας. Σε μεγάλη κλίμακα έχουμε επενδύσεις που δόθηκαν μέσω των διαφόρων μέσων ανάμειξη χρηματοδοτήσεω από το 2007 μέχρι το 2015. Είχαμε πολλά προγράμματα, 112 ενεργειακά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν με πολλά αποτελέσματα. Φέτος, αρχές του έτους, ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία Electrify για ηλεκτροδότηση και εκεί συμμετέχουν μικροί ιδιωτικοί επενδυτές και είχαμε αρχικά μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αρχές του έτους. Καταπληκτικά αποτελέσματα. 190 ε, προτάσεις λάβαμε από μικρές επιχειρήσεις αναλύουμε τις προτάσεις για να δούμε τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ήταν επιτυχές το πρόγραμμα ηλεκτροδότησης, όχι μόνο ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά προσελκύσαμε και άλλους εταίρους στην Αφρική, στη ΣΥΠΑ. Δέκα εκατομμύρια ε, δολάρια δόθηκαν από τους εταίρους για τις επενδύσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε θετικό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. Να αποφευθεί η διαφθορά, να δημιουργήσουμε καλύτερο περιβάλλον. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τεχνική ε, αρρωγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε να στείλουμε τάχιστα εμπειρογνώμονες να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τους εταίρους, να βοηθήσουν τον κόσμο, τους ντόπιου να δημιουργήσουν ε, δυναμικό, να τους δώσουμε συμβουλές για τα διάφορα προγράμματα ηλεκτροδοτήσεως. Το σημαντικότερο είναι να αισθανθούν τα κράτη όταν στερνίζονται την πολιτική, ότι είναι δική τους. Το είπατε και στην αρχή. Έχουμε 30 χώρες που έχουν εστιάσει την προσοχή τους στον ενεργειακό τομέα, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω διαλόγου και μέσω κοινών διακηρύξεων με 19 χώρες για διαβριμένη συνεργασία για την ενέργεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνεργασία με τις χώρες αυτές. Να είναι στο επίκεντρο της προσοχής οι κυβερνήσεις, χωρίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς την κατάλληλη πολιτική, χωρίς το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι κυβερνήσεις για να γίνουν μεταρρυθμίσεις, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τέλος, εξίσου σημαντικό, εκτιμούμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Να επενθυμίσω ότι έχουμε διάφορα προγράμματα για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για την εκτροδότηση της υπαίθρου, κυρίως στις λιγότερο ενεπτυγμένες χώρες. Και το θέμα του φίλου επίσης σημαντικό. Εφαρμόζουμε θεματολόγιο ε, ενεργειακό ηλεκτροδοτήσεως για να στηρίξουμε τις γυναίκες να βοηθήσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες, να τις στηρίξουμε όταν έχουν προγράμματα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Καλύπτουμε σφαιρικά τα θέματα αυτά. Λαμβάνουμε υπόψη και τα επιτεύγματα και τα προβλήματα μετά την COP21. Τις δεσμεύσεις του αναλήφθησαν σε επίπεδο COP21 κυρίως ε, έχοντας σαν στόχο την καταπολέμηση των αποτελεσμάτων τη αλλαγή του κλίματος. Ευχαριστώ που μας ενημερώσατε όσον αφορά το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόλι έχει το λόγο για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πάρα πολλά στα σχόλιά σα, Θα ήθελα σε πολλά να απαντήσω. Ίσως μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε λεπτομέρειε. Κάτι να επαναλάβω πολύ σωστά αυτά που είπατε, πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Πρέπει να συνεχίσουμε και το τονίζω. Επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο αυτές οι κοινότητες. Μπορεί να γίνει προσβάσιμο το δίκτυο αν υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης. Αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα. Δεν είναι επιλογή μεταξύ δύο πραγμάτων Θέλουμε πάντα να ξεκινήσουμε με αποκέντρωση. Αυτή είναι η σωστή αρχή. Όταν μιλάμε για απόμακρε κοινότητε τη υπαίθρου. Τώρα για, για το βιολογικό αέριο, βιοαέριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολλές από τις κοινότητες που αναφέραμε βασίζονται στη γεωργία. Πολλοί ενδιαφέρον και βιώσιμος τρόπος να χρησιμοποιήσουν τα απόβλητα των εκμεταλλεύσεων. Ίσως μετά από ε, το θερισμό, μετά τη συγκομιδή, ε, τα απόβλητα των ζώων, κυκλική οικονομία. Έχω, αν έχουμε μια γεωργική κοινωνία, που πολλές από αυτές είναι γεωργικές αγροτικές οικονομίες ή αλληλευτικές κοινωνίες, περίπου, μπορεί να καλυφθούν από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση ε, μιλάμε περισσότερο για τη συντήρηση των ε, αλλιευμάτων. Για τους παραγωγούς, εκείνους που ζουν στα χωριά και παράγουν διάφορα βασικά προϊόντα. Χρειάζεται να μπορούν να συντηρούν τα προϊόντα τους. Να τους βρούμε έναν τρόπο να τα συντηρούν, να τα πηγαίνουν στην αγορά τη σωστή στιγμή, για να παίρνουν και την καλύτερη τιμή για τα αγαθά τους. Γιατί δούλεψαν και σκληρά για να παράξουν αυτά τα προϊόντα. Ίσως εκεί θα ήθελα να κλείσω και να ολοκληρώσω τα σχόλιά μου, ευχαριστώντας σας για τα σχόλια τα δικά σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είδατε από την ανταπόκριση συναδέλφων πόσο εξετίμησαν τη δουλειά που κάνετε, πόσο εκτιμούν τη δουλειά σας και προσβλέπουν τη συνεργασία μαζί σας. Έχετε τις πληροφορίες, ε, όνομα, τηλέφωνα κλπ. Έχετε λεπτομέρειες, email, διεύθυνση email Ευχαριστούμε όλοι που ήρθε σήμερα. Πολύ έξοχη ήταν η παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Α, να πω κάτι. Ξέχασα. Έχουμε προφορική ερώτηση. Σχέδιο ψηφίσματος μάλλον. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και για τα δύο Παρασκευή 14 Οκτωβρίου το μεσημέρι στις 12. Συνάδελφοι, εδώ συμφωνούμε σχετικά με πρέπει να συμβεί. Ίσως οι ομάδες μπορούν να συνεργαστούν ούτω ώστε τα μηνύματα του ψηφίσματο να είναι σαφή. Δεν έχουμε πολλέ τροπολογίε που να επαναλαμβάνονται και να κολλάνε σε λέξει. Να έχουμε 9 ή 10 σαφεί συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε ότι είναι ανοιχτή. Θέλουν να επεξεργαστούν τα θέματα. Αν μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε γι' αυτό, πριν ψηφίσουμε, να είμαστε σίγουροι για ότι θα κάνουμε συμβιβασμού για να βγει ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι ένα μακροσκελέ κείμενο με θολό μήνυμα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 9 τώρα της ημερήσιας διατάξης. Oh, Εντάξει, συνάδελφοι, περάσουμε στο σημείο 9. Βασικά, πριν από αυτό, θα να πω ότι από ό,τι είδα, μόνο ένα θα είναι το θέμα της ψηφοφορία αύριο το πρωί. Αντί να ξεκινήσουμε στι 9, προτείνω να ξεκινήσουμε στις 9 και μισή. Εντάξει, συμφωνείτε όλοι και συντονιστέ. Αν μπορεί να τη το μήνυμα και η γραμματεία ότι θα ξεκινήσει στις 9.30 αύριο η συνεδρίαση, θα κάνουμε τη ψηφοφορία και μετά στις 10 ε, θα πάμε στην άλλη αίθουσα ε, για να συνεδριάσουμε μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. 9.30 λοιπόν αύριο. Θα ενημερωθούν και οι συνάδελφοι και όχι μόνο μέσω mail. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο ε, για την ε, αποστολή παρακολούθηση των εκλογών ε, στη Ζάμπια. Η κυρία Κέγκε δεν έχει φτάσει ακόμα γιατί υπήρχε καθυστέρηση στην πτήση και ο Μάικλ ήταν επικεφαλής της ομάδας, δεν είναι εδώ, όμως έχουμε ένα άλλο μέλος εδώ της αντιπροσωπείας και εγώ ξέρω ότι πήγαν καλά τα πράγματα σε εκλογές ε, ειρηνικά, όμως υπήρχαν ε, κάποια ζητήματα. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση στην Αφρική σε αυτό το πεδίο σε πολλές χώρες, ε, οπότε δεν ξέρω, μπορείτε να μας πείτε κι εσείς τι συμβαίνει με τη Ζάμπια, παρακαλώ. Thank you. And, um, I'm hoping Cecile arrives so that she can answer all the difficult questions, because um, as you heard, I was just part of the uh, smaller parliamentary observation group. So when... Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε μια φωτογραφία σχετικά με αυτά που συμβαίνουν. Ακουγόμαστε καθαρά από την ελληνική καμπίνα. Θα είχα την καλωσία μα κάνετε ένα ανέβημα προ την καμπίνα υπαριθμών 7. Μα ακούτε καθαρά.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 δεν χαρακτηρίζεται η χώρα από αυτό. Ελπίζαμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό. Και το τονίζαμε αυτό. Εκφράζαμε ανησυχίες εκείνη για τα τεκτενόμενα. Και ελπίζαμε ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί. την ίδια μέρα έγιναν πέντε ψηφοφορίε. Προεδρικέ κοινοβουλευτικέ και άλλε. Και ένα δημοψήφισμα. Που δεν πέρασε το κατάλληλο όριο. Και οργανώθηκε τελευταία στιγμή. Το UPND, το κυρίαρχο κόμμα, ζήτησε από τους υποστηριχτές του να υποκοτάρουν την ψηφοφορία. Έγινε μεγάλη μάχη για τι προεδρικέ. Είχαν γίνει και άλλε πριν από 15 μήνες προεδρικέ. Υπήρχε διαφορά με 28.000-38.000 ψήφους. Πολύ μικρή διαφορά στις προηγούμενε εκλογές. Ήταν σχεδόν ε, εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Σκληρή μάχη λοιπόν για τι προεδρικές πριν από 15 μήνες. Είχαμε 9 υποψηφίους για πρόεδρο. Η διαφορά ήταν μικρή. Δικοματική ήταν η μάχη. Είχαν καινούριο εκλογικό νόμο πρόσφατα. Έπρεπε να έχει 50% ε, των, των ψηφοφόρων εκείνος που νίκουσε. 50 συν 1 για να νικήσει κάποιο αλλιώς γινόταν, προβλεπόταν δεύτερος γύρος. θα ήξερε ο κόσμος όλα αυτά, στα εκλογικά τμήματα, όταν γινόταν η καταμέτρηση. Βλέπαμε λοιπόν ότι γίνεται μάχη στήθος με στήθος. 50,35% πήρε ο πρόεδρος. Άρα πολύ μικρή διαφορά. Μικρές οι διαφορές λοιπόν μεταξύ των υποψηφίων. Τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Στην αρχική μας έκθεση τα έχουμε συμπεριλάβει όλα αυτά τα ζητήματα. και οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο όταν υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των υποψηφίων την ημέρα των εκλογών. Όλα πήγαν καλά, ήταν καλά οργανωμένα. Επικρατούν μεγάλες ανισότητες στη χώρα. 20% του πληθυσμού έχουν ηλεκτρική ενέργεια στα εκλογικά τμήματα η μέτρηση γινόταν με το φως του ηλίου και με λάμπες πετρελαίου κλπ. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Και οι υπεύθυνοι για την καταμέτρηση των ψήφων είχαν πάει την προηγούμενη νύχτα και κοιμηθήκαν στο εκλογικό τμήμα, να είναι εκεί να μετράνε την άλλη μέρα. διεξήχθησαν ειρηνικά οι εκλογές. Ήταν υπομονετικοί οι πολίτες. Και έκαναν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε να ψηφίσουν. Και το προσωπικό στα εκλογικά τμήματα ήταν πολύ επαγγελματικό. Ήταν μακροσκελής η διαδικασία στην ημέρα των εκλογών. Οι εκλογικοί κατάλογοι έφτασαν καθυστερημένα. Οι παρατηρητές ήταν στα εκλογικά τμήματα. Ανήκαν σε πολιτικά κόμματα, στην κοινωνία των πολιτών. Έμπαινε κανείς, έδειχνε την κάρτα του. Γινόταν τα δέοντα, οι ελεγκτές έλεγχαν αν υπάρχει ωστή αντιστοιχεία ταυτότητας και μετά πήγαινε ο ψηφοφόρος να πάρει τα πέντε ψηφοδέλτια και να πάει να ψηφίσει. Ήταν αργοκίνητη διαδικασία που θα μπορούσε να επιταχυνθεί. Κάποιοι άνθρωποι είχαν πάει δύο-τρεις ώρες πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα. και οι ουρές κρατούσαν επί μακρόν διότι ήταν αργή όλη η διαδικασία. Παρόλο που οι υπάλληλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Άρα κάτι γινόταν, τα προσπάθεια. Η καταμέτρηση των ψήφων ήταν δυσχερής. Την προτιμωσία για τις εκλογές όσο συνέβησαν καθοδόν προς τις εκλογές έπαιξαν περισσότερο ρόλο από αυτά που διαδραματίστηκαν την ημέρα των εκλογών αυτή καθε αυτή. Η κυρία Αγκέγγι αναφέρθηκε σε διάφορα στοιχεία που αφορούν τις εκλογές ή θα τα πει όταν έρθει. Το θέμα που ετέθη ήταν η ελευθεροτυπία, ο περιορισμός των ΜΜΕ, η αμεροληψία των ΜΜΕ, η ο κρατικός σταθμός υποτίθεται ότι θα ήταν αμερόληπτος. Εμείς διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αμεροληπτικά τα κρατικά μέσα. Στήριζαν το κυβερνόν κόμμα και τον πρόεδρο. Όσον αφορά την κάλυψη των εκλογών, και διάφοροι δίσκου που παρουσιάζαν, προωθούσαν τον πρόεδρο καλύπταν πολύ περισσότερο τον πρόεδρο από ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαν κλείσει κάποιες εφημερίδες πριν λόγω μη καταβολής φόρων, ούτως πίν. Άρα τα ΜΜΕ δεν ήταν αμερόληπτα. Δεν υπήρχε ρύθμιση για τα εκλογικά μηνύματα των διαφόρων κομμάτων και την ε, διάθεση του χρόνου και του χώρου. Είχαμε πολιτική διαφήμιση που παρουσιαζόταν και παρουσιαζόταν πριν ένα μήνυμα της Επιτροπής των Εκλογών και δεν ήταν σαφή τα όρια μεταξύ των διαφόρων μηνυμάτων που παρουσιαζόταν στα ΜΜΕ. Άρα, ελευθερία των ΜΜΕ, αμεροληψία των ΜΜΕ, τα σοβαρά θέματα. Οι διατάξει για τη δημόσια τάξη. Και η εκστρατεία υπέρ του Προέδρου. Αν πήγαινε σε εκστρατεία Προέδρου σε μια επαρχία συγκεκριμένη, η αντιπολίτευση δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο ακυρώθηκαν κάποιες συγκεντρώσεις την τελευταία στιγμή γι' αυτό το λόγο. Και λόγω του μεγέθους των επαρχιών αποκλειόταν να συναντηθούν ή να συμπέσουν τοπικά οι δύο συγκεντρώσεις. Άρα ήταν, εξετάσαμε το ρόλο που έπαιζε ο, ο πρόεδρος και αυτοί που τον υποστήριζαν εν συγκρίση με την υποστήριξη που παρεχόταν από τα ΜΜΕ στους αντιπάλους. Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Εκλογών έκανε αρκετά καλή δουλειά κατά την άποψή μας, ετύχανε εμπιστοσύνη. Τα μέλη αυτής μπορούν να απολυθούν από τον Πρόεδρο και αυτό ίσως βοηθήσει στο μέλλον να επιτευχθεί η αμεροληψία της Ανλόγου Επιτροπής. Αμφισβητήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα. Έχει ανακηρυχθεί ο πρόεδρος, έχει αναλάβει τα καθήκοντά του. Ελπίζουμε αυτά τα σποραδικά επεισόδια συγκρούσεων να μην συνεχιστούν στο μέλλον. Πρέπει να αισθανθεί ο λαός ότι έχει λόγο έγιναν ταυτόχρονα οι εκλογές την ίδια μέρα για διάφορα, διάφορες, ε, διάφορα αξιώματα. Αυτά ήταν έτσι σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η εικόνα των εκλογών, πάρα πολύ σύντομα, τι έγινε. Μια φωτογραφία, ευχαριστώ για τη φωτογραφία, μας δίνει μια σαφέστατη εικόνα, λέει πρόεδρος. Μιλήσαμε πρόσφατα στην ενέργεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Και δεν είχα σκεφτεί τι κάνει κανεί με τη διεξαγωγή των εκλογών. Άμα δει ο ήλιος, τι κάνεις. Κλείνεις το εκλογικό τμήμα, δεν έχεις φως. Πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ενέργεια. Πρέπει οι συντονιστές ίσως να το θέσουν σαν προτεραιότητα τον επόμενο χρόνο. Να έχουμε υπόψη μα τα χωριά που είναι εκτό δικτύου. Αυτό συζητάγαμε πριν έρθετε. Οι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν ερώτημα στη Τζιν. Θέλουν να μιλήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Λάτε Κόλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Ο κύριος Κόλ θα μιλήσει εκ μέρους της ε, Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης για τις εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ αξιότιμα μέλη που έχετε θέσει αυτό το σημείο στη διάταξη. Θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα έχει ήδη αναφέρει η κυρία Λάμπερτ. Πράγματι, βρισκόμαστε στα τελικά στάδια αξιολόγηση τη εκλογική διαδικασία. Επομένω, ακόμα εκπονείται τελική έκθεση και θα προετοιμαστεί για την επαναληπτική επίσκεψη τη επικεφαλή τη κυρία Κιάνγκε που ελπίζουμε να λάβει χώρα το πρώτο ίνιση του Νοεμβρίου όπου το πιο σημαντικό είναι ότι θα παρουσιάσουμε τις ε, κύριες συστάσεις που έχουμε ε, αναπτύξει ε, υπόψη των αξιωματούχων της Ζάμπια. Ενώ η Εκλογική Επιτροπή έδειξε επαγγελματισμό στις προετοιμασίες της και παρά ζητήματα έλψης εμπιστοσύνη και ε, κατηγορίες ε, για μεροληψία σε συγκεκριμένα σημεία. Πολλά ενδιαφέροντα μέρη εξέφρασαν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, η διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία δεν ήταν τέλεια και σε κάποια ε, κέρια ζητήματα καταμέτρησης ψήφων Εκεί θεωρούμε ότι χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες επειδή δεν δόθηκε πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων στα εκλογικά κέντρα παρά τα πολυάριθμα τέτοια αιτήματα. Και λόγω της ε, συνεχιζόμενης αποσταθεροποίησης θεωρούμε ότι η ενίσχυση τη αξιοπιστία, της εκλογική διαδικασίας ε, δεν επετεύχθη όσο θα θέλαμε. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η εκστρατεία ήταν ε, αρκετά καλή για τα δεδομένα της περιφέρειας, ωστόσο οι ίδιοι οι Ζαμπιανοί θεωρούσαν ότι ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα επιθετική. Είχαμε το λυπηρό περιστατικό του θανάτου ενός ε, από τους ε, υποστηρικτές. Εξαιτία ε, τη καταστολή από τι αστυνομικέ δυνάμει που οδήγησε σε αναστολή τη εκτρατεία σε μεγάλο μέρο τη Λουσάκα, αλλά όχι μόνο. Θεωρούμε ότι αυτό δείχνει έλλειψη ετοιμότητας ε, των αστυνομικών αρχών να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, συγκεντρώσεις πολιτών με μη βίαιο τρόπο. Στις 22 Αυγούστου είχαμε αυτή την αναστολή λοιπόν. Ακριβώς μετά τις εκλογές όταν υπευλήθη η έφεση ε, και καταγγελία των εκλογικών αποτελεσμάτων, το οποίο ήταν λυπηρό, όταν λοιπόν ανεστάλησαν οι άδειες τριών ε, ε τηλεοπτικών μέσων το Movie TV, το μοναδικό κανάλι που δεν ήταν ανοιχτά υπέρ τη κυβέρνηση και είχαμε και δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, των οποίων οι άδειε ανεστάλησαν. Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία έκφρασης. Η μοναδική εφημερίδα υπέρ της αντιπολίτευσης έχει πληγεί πολύ σημαντικά, μάλλον έχει ε, σταματήσει η κυκλοφορία της ε, για υποτιθέμενους ε, φόρους που ακόμα χρωστά εφημερίδα. Και υπάρχουν διφορούμενες απόψεις και όλα αυτά τέλος πάντων έχουν επιδράσει αρνητικά στην ενημέρωση των πολιτών. Κάτι άλλο το οποίο προέκυψε σαφώς από την αξιολόγησή μας είναι ότι το πατριωτικό μέτωπο ε, ε, εποφελήθηκε υπερβολικά από τη θέση του. Υπήρξαν συγκεκριμένες ελλείψεις ε, σε σύνδεση με την χρηματοδότηση και αυτό οδήγησε σε μη ισοπεδίο ανταγωνισμού για όλα τα κόμματα. Ήταν ε, πολύ κοντά τα αποτελέσματα, 50,35% των ψήφων υπέρ του Πρέδρου Λούγκου. Με πολύ μικρή πλειοψηφία λοιπόν πέρασε το 50 που είναι η προπόθεση για να εκλεγεί κανείς. Το κόμμα της αντιπολίτευσης υπέβαλε ένσταση στο αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρου στις 19 Αυγούστου, ζήτησε από το Σταγματικό Δικαστήριο να ε, αποφανθεί ότι δεν εξελέγει νόμιμα ο υποψήφιος και ότι έτσι ήταν άκυρο το αποτέλεσμα, λόγω μη συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο. Η αίτηση βασιζόταν κυρίως σε επιχειρήματα που αφορούσαν το εκλογικό περιβάλλον, μεροληψία για παράδειγμα στα μέσα ενημέρωσης, περιορισμοί ε, στην ε, κυκλοφορία και εκστρατεία άλλων πολιτικών κομμάτων, καθώς και υποτιθέμενες ε, παρατυπίες σε ό,τι αφορά ε, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την καταμέτρηση, αλλά και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ε, απερίφθη η αίτηση ένστασης αυτή για διαδικαστικούς και κυρίως λόγους. Τρεις με δύο ήταν η απόφαση. Απεφάνει το δικαστήριο ότι δεν είχε το δικαίωμα να παρατείνει το διάστημα 14 ημερών που ε, ήταν απαραίτητο για την ακροματική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ένσταση. Αυτά από πλευρά μα. Έχετε και πάλι το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Σεσίλ. Ξέρω ότι είχε καθυστέρηση η πτήση σου. Πάνω που θα σου έστειλα ένα μήνυμα να μην βιάζεσαι, γιατί είχαμε μια πολύ καλή έκθεση και αναφορά από την κυρία Λάμπερτ, αλλά και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Παρακαλώ. Θα μιλήσω Ιταλικά αφού υπάρχει διερμηνία. Ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω. σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ζάμπια. Από τέλος Ιουνίου ε, μέχρι Σεπτέμβριο ε, ανεβλήθη αυτή. Είχαμε από 28 κράτη-μέλη παρατηρητές συμπεριλαμβανομένης Νορβηγίας. Θέλω να αξιολογήσουμε την όλη διαδικασία σύμφωνα τα διεθνή πρότυπα για διαφανείς και ειλικρινείς εκλογές. Στις 11 Αυγούστου έγιναν εκλογές. Ήταν πρόκληση, πολύ μεγάλη, για μια χώρα όπως η Ζάμπια. Πρώτες που έγιναν σύμφωνα με το νέο σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο. Ο αριθμός των εδρών αυξήθηκε και σημαντικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εκλογική επιτροπή έπρεπε να διοργανώσει την ψηφοφορία και πέντε ε, ψηφοδέλτια. Την ημέρα των εκλογών παρακολουθήσαμε την ψηφοφορία και την καταμέτρηση σε 520 εκλογικά τμήματα και στις 10 επαρχίες. Το αποτέλεσμα αξιολογήθηκε θετικά. Θετικό από τα, στα, 97% των εκλογικών τμήματων. Ακολουθήθηκαν σωστές διαδικασίες καταμέτρησης. Υπήρχαν αναγκαίες εγγύσεις για την ακαιρεότητα της ψηφοφορίας και για την πρόσβαση στην ψηφοφορία. Για του εκλογικού ελέγχου υπήρχε κατάλληλο προσωπικό. Όμως το προσωπικό για τον έλεγχο μέτρηση των ε, εκλογικών τμήματων δεν εξακρίβωναν κατά πόσο έβαζαν ε, ανεξίτηλο μελάνι στα δάχτυλα των ψηφοφόρων. Και δεν γινόταν σωστή, ε, σωστός έλεγχος των ψηφοδελτίων πάντα. Η μέτρηση των ψηφοδελτίων έγινε σωστά. Τέσσερι εκλογέ και ένα δημοψήφισμα έγινε και την ημέρα. Το πέμπτο, ε, η πέμπτη συμφορία ήταν δημοψήφισμα. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια διοργάνωσης και ευαισθητοποίηση των εκλογέων. Υπήρξαν κάποιες αδυναμίες. Η Επιτροπή διοργάνωση των Εκλογών στη Ζάμπια έδειξε επαγγελματισμό. Παρά τι αρχικέ καχυποψίες και κατηγορίες περιμένων ψίες από την αντιπολίτευση. Τελικά, δημιουργήθηκε κλίμα εμπιστοσύνη όσον αφορά τις εκλογές. Η Επιτροπή έκανε προσπάθειες για αύξηση της διαφάνειας. Κάτι σημαντικό. Δεν επέτρεψε ούτε στους παρατηρητές τους διεθνείς, ούτε στους εθνικούς πρόσβαση σε διάφορες εκλογικές αστεριότητες χάθηκε η δυνατότητα να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στις εκλογέ. Η, η, η, εκλογική αυτή επιτροπή δεν επέτρεψε να έχουν πρόσβαση στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων στα κέντρα κατά μέτρης εθνικά. Και αυτό παρά τις προσπάθειές μας για πρόσβαση. Χάσαν έτσι μια ευκαιρία να ενισχύσουν περαιτέρω την αξιοπιστία των εκλογών. Κάποιες δηλώσεις από το πατριωτικό μέτωπο και από το Ενωτικό Κόμμα για την ε, Εθνική Ανάπτυξη, το UPND, αύξησαν τις εντάσεις στη χώρα. Η διακοπή της εκστρατείας στη Λουζάκα και στην Αμουάλα, τη νότια αυτή επαρχία, επηρέωσε τα μικρά ε, κόμματα και κάποιους ανεξάρτητους υποψηφίους. Οι δυνάμεις της τάξης έκαναν προσπάθειες για την τάξη. Κινήθηκαν καλύτερα οι δυνάμεις της τάξης σε κάποιες επαρχίες και λιγότερο καλά σε άλλες. Δεν υπήρξε ισοτιμία όσον αφορά την κάλυψη των εκλογών. Άρα δεν μπορούσαν καλά πληροφορωμένοι οι εκλογείς. Στηρίχθηκε κυρίως το κυβερνών κόμμα στα ΜΜΕ. το δεπόστ, το έντυπο, το ιδιωτικό ε, περιορίστηκε. Άρα μειώθηκε η ελευθεροτυπία. Και το αναφέραμε αυτό. Η αντιπολίτευση δεν είχε την ίδια πρόσβαση στον έντυπο τύπο. Στις 22 Αυγούστου η ανεξάρτητη αρχή για τα ΜΜΕ διέκοψε το μοναδικό κανάλι τηλεόρασης, το Movie TV, που ήταν ιδιωτικό κανάλι και δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εσιώπησε. Αυτό έχει αρνητική α, συνέπεια στη ροή των πληροφοριών σε πολύ ευαίσθητη περίοδο των, των εκλογών. Η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου ήταν κάτι καλό για τις εκλογές. Όμως εφαρμόστηκε το Public Order Act. Περιορίζονται τις δυνατότητες συγκέντρωσης των ανθρώπων κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κυβερνών κόμμα ευνοήθηκε από τη θέση του. Και παρατηρήσαμε ότι η χρήση των κρατικών πόρων για εκλογικούς σκοπούς παραβίαζε τον νόμο και συνέβαλε σαν ισότητα των συνθήκων μεταξύ των διαφόρων στρατοπέδων. 15 Αυγούστου, η Εκλογική Επιτροπή της χώρας ανακοίνωσε τελικά αποτελέσματα των προεδρικών. Ο πρόεδρος Λούγκου του PF με 1867 ψήφους εξελέγει διότι είχε 50,35% ε, των ψήφων ξεπερνώντας κατά λίγο το 50% που είναι το όριο για να εκλεγεί πρόεδρος κανείς. Υποψήφιος του UPND, Σιλέμα, είχε 1.760 ψήφους. 347. 47,63% από τις ε, ψήφους. 100.530 ψήφοι ήταν η διαφορά. Οι υπόλοιποι ψήφοι πήγαν στα άλλα κόμματα. Η ψηφίος η Τσιλέμα του UPND έκανε ένσταση για τα αποτελέσματα αμέσως μετά τις εκλογές. Έκανε προσφυγή λοιπόν. Υπέβαλε ένσταση και ζήτησε το συνταγματικό δικαστήριο να ακυρώσει τι εκλογέ. Διότι δεν έγινε σεβαστό το νομικό πλαίσιο των εκλογών. Απερίφθη η ένσταση στις 5 Σεπτεμβρίου χωρί δυνατότητα προσφυγή Μετά με απόφαση του δικαστηρίου που δηλώνει ότι το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να παρατείνει συνταγματική περίοδο για ακροάσεις κατά 14 μέρες. Είχε εκπνεύσει 2 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα να μπορεί το εκπρόσωπος αντιπολίτευσης να πάει να εισακουστεί. δημιουργήθηκαν προβλήματα. Δύο δικαστέ ε, ξέφρασαν διαφορετική άποψη σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου. Κλείνοντα. να πω ότι οι περισσότερε 14 μέρε αφορούσαν προδικαστικά θέματα. Το δικαστήριο δεν κατέφερε να δώσει σαφή απόφαση. Εγκαίρω, σύμφωνα με τις προθεσμίες προβλέπονται. Άρα οι υποβάλλοντας την ένσταση δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω δημόσιας ακρόασης. Άρα υπονομεύθηκε η εμπιστοσύνη στο μηχανισμό προσφυγής κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών. Εδώ έγκυται και η αδυναμία της διαδικασίας, το αναφέρω στην έκθεσή μου. Παρακολουθήσαμε τα πάντα και αυτό το αναφέρουμε και στις συστάσεις που κάναμε μετά την παρατήρηση των εκλογών. Ναι, θα ήθελα να δώσω κάποιες... Σας ευχαριστούμε που δώσατε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, θα σας ακούσαμε. Θέλει κάποιος συνάδελφος να υποβάλει κάποια πρόσθετη ερώτηση. Εάν όχι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομιλήτρια για την παρουσίαση της παρόλο που υπήρχε αυτή η καθυστέρηση στη πτήση της. Θα συνεχίσει η υποστήριξή μας προς τη Ζάμπια, γιατί τώρα πλέον δεν θα κάνουμε μια απλή παρατήρηση των εκλογική διαδικασίας, αλλά θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγι στις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα. Συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 9.30 έχουμε την ψηφοφορία αύριο και στις 10 θα αλλάξουμε αίθουσα, θα πάμε στο 2Q2 για να συνδέσουμε και από με την ΑΦΕΤ. Και θα ήθελα επίση να του συναδέλφους στις 6.30 στο δεύτερο όροφο, έναν όροφο κάτω από την Ολομέλεια, θα υπάρξει φωτογραφική έκθεση για την ε, Ανατολική Αφρική. Εγώ οπωσδήποτε θα δω αυτή την έκθεση στις 6.30, σε μισή ώρα. Ευχαριστώ συνάδελφοι.